Buenos días. Καλημέρα σας. Σε αυτή την ε, γκρίζα ημέρα στις Βρυξέλλες, ε, σε αυτή την αίθουσα θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Ας έχουμε κάποια δυναμική, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα να προσεγγίσουμε στη μέση και λίγο χρόνο. Δύο ανακοινώσει το βραβείο Ζαχάροφ ε, για την ελευθερία έκφρασης και σκέψης ε, στις 29 ε, Οκτωβρίου Οκτωβρίου αποφασίστηκε σε ποιον θα δοθεί. Θα γίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 16 Δεκεμβρίου μία εκδήλωση και θα παραδοθεί τον ε, βραβείο στο Ραΐφ Μπαντάουι πιστεύω ότι θα υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αντίκτυπος στις 16 Δεκεμβρίου με την απονομή αυτού του βραβείου. Βέβαια, υποθέτω ότι ο κ. Μπεντέρου δεν θα μπορέσει να το παραλάβει. Αλλά ελπίζω ότι η γυναίκα του και τα παιδιά του να μπορέσουν να μετακινηθούν στο Στρασβούργο. Να σας ανακοινώσω επίσης ότι στις 3 Δεκεμβρίου στις 11.30 μια επίσημη αντιπροσωπεία του Εθνικού Κογκρέσου του Κινέζικου Λαού. Κύριε Πρέντε, γιατί καθίσατε τόσο μακριά. Ελάτε εδώ δίπλα. Φαίνεται λες και έχουμε τσακωθεί. Πλησιάστε. Γιατί πήγατε εκεί και καθίσατε ολομόναχος τόσο μακριά. Λοιπόν, στις 3 Δεκεμβρίου, στις 11.30, όπως σας είπα, θα συναντηθούμε με εκπροσώπους ε, του Εθνικού Κινέζικου Κογκρέσου και όλοι οι συνάδελφοι από αυτή την υποβιτροπή είναι προσκεκλημένοι για να κάνουμε μια συζήτηση για το Θιβέτ. Και τώρα έχουμε εδώ τον κύριο Πρέτα που ήρθε και δίπλα μας και θα δούμε την ε, ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο, το 2014 και την πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση επί του Θέματο και τι σχετικέ τροπολογίε. Θα δώσω λοιπόν κατευθείαν το λόγο στον κύριο Πρέντα. Θα ήθελα να το συγχαρώ γιατί και ο ίδιος αλλά και όλοι οι σκιώδεις συζητητές συνεργάστηκαν πολύ καλά και θα ήθελα να επενθυμίσω ότι προβλέπεται η ψηφοφορία στην ΑΦΕΤ στις 16 Νοεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Κύριε Πρέντα, έχετε το λόγο. Euh, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Βεβαίως η ψηφοφορία προβλέπεται για τη Δευτέρα και θα ήθελα να πω ότι όπως κάθε χρόνο αυτή η έκθεση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον ε, στα μέλη της Επιτροπής μας και και για τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων έχουμε λάβει 420 τροπολογίες, δεν είναι άσχημα. Και όπως ανέφερα στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων, εδώ και 1,5 μήνα, θεωρώ ότι θα ήταν σημαντικό από την άποψη της μορφής του τύπου αυτής της έκθεσης να είναι σύντομη έκθεση, να είναι συνοπτική. Είχα εξηγήσει τότε ότι η αναγνωσιμότητα της έκθεσης είναι κάτι το σημαντικό και για το λόγο αυτό πρότεινα 48 τροπολογίες συμβιβαστικές ένας αριθμός ε, λοιπόν ικανοποιητικός τροπολογιών και προσπάθησα έτσι να μειώσω όσο το δυνατόν περισσότερο τις επαναλήψεις, τις πλεονάζουσες επαναλήψεις, εφόσον ζητούμε από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων να συντάξει μια έκθεση για την πολιτική ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία που να είναι αναγνώσιμη. Δεν μπορούμε λοιπόν εμείς να πράττουμε το αντίθετο. Αυτή είναι η ιδέα. Και εξάλλου ανησυχώ λίγο διότι ε, μου είπαν ότι στην Επιτροπή Γυναικών θα υπάρξουν περίπου 60 παράγραφοι. 60 παράγραφοι. Είναι κάτι από μία επιτροπή, είναι πολύ. Είναι πάρα πολύ ψήφισα πριν από δύο μέρες στην Επιτροπή ΔΕΒ. 12, ε, ε, είναι 12 παράγραφοι εκεί σε αυτή την Επιτροπή. Λοιπόν, κάνω έκκληση, δεν ξέρω αν υπάρχει εδώ κάποιος από την Επιτροπή Γυναικών, αλλά 60 παράγραφοι, δεν πρέπει κανείς να υπερβάλλει. Μπορεί αυτές οι 60 παράγραφοι να ε, είναι πιο ογκώδεις από την ίδια μου την έκθεση. Ξέρω ότι τα θέματα των γυναικών είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ελπίζω ότι θα έχουμε στο τέλος κάτι το οποίο να είναι χρησιμοποιήσιμο. Και για να επανέλθω στις 420 τροπολογίες, όταν έλεγα ότι, είχαμε, ότι έχουμε 48 συμβιβαστικές τροπολογίες και είχαμε συνεδριάσει στο Στρασβούργο, επί της ουσίας και διαβουλεύσεις γραπτές. Και πρέπει να ομολογήσω ότι είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία με τον εισηγητή, τον σκιώδη εισηγητή, τους σκιώδης εισηγητές όλων των πολιτικών ομάδων και νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι καλό για όλες τις πολιτικές ομάδες. Ο καθένας έρχεται με τη δική του προοπτική εικόνα από την ομάδα του, αλλά νομίζω ότι ο συμβιβασμός είναι ένας καλός συμβιβασμός για όλους μας. Εφόσον και οι τροπολογίες C48 αναφέρονται σε σημαντικό αριθμό θεμάτων, ε, για τα οποία θέματα η Επιτροπή αποδίδει ιδιαίτερη σημασία και με αυτές τις συμβιβαστικές τροπολογίες συμφωνήσαμε να επισύρουμε την, αν, την προσοχή πάνω στην ανάγκη να υπάρχει μια ε, συνεκτικότητα ανάμεσα στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική της Ένωσης και συμφωνήσαμε ότι η Ένωση θα πρέπει να επιμείνει πάνω στην υλοποίηση της πολιτικής ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία για να βελτιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα των μέσων αυτής της πολιτικής και θα ήθελα να συγχαρώ για το διάλογο, για τις στρατηγικές αναχώρα και έχουμε τον ειδικό εκπρόσωπο ε, για το ενδιαφέρον αυτό θέμα και τον συγχαίρω έπρεπε να συνεχίζουμε με τις εξωτερικές πολιτικές να προωθούμε τα δικαιώματα. Πρόκειται για την πολιτική διεύρυνσης, γειτονίας και ανάπτυξης και για την εμπορική πολιτική. Αυτό περνάει επίσης από μια διαχείριση που να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και που να σέβεται την εξωτερική διάσταση της κρίσης των προσφύγων που προσπαθούν να έλθουν στην Ευρώπη. Συμφωνώ και είμαι ικανοποιημένος επειδή τη βρήκαμε μια κοινή γλώσσα για το θέμα αυτό. Ε, έχουμε βεβαίως εδώ δεν θα επιλύσουμε αυτό το θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ περίπλοκο δεν έπρεπε λοιπόν να μεταμορφώσουμε αυτή την έκθεση σε μια έκθεση που αναφέρεται μόνο ε, στο θέμα της μετανάστευσης. Νομίζω ότι βρήκαμε μια κοινή γλώσσα για το θέμα αυτό. Ο συμβιβασμός αφορά με την εμπορία ανθρωπίνων όντων, ε, με την ε, θανατική ποινή, με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και για τα δικαιώματα του παιδιού και της γυναίκας συμφωνήσαμε για την σημασία να κρούσουμε τον κόδανα του κινδύνου για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, διότι η κοινωνία των πολιτών έχει γίνει εύθραυστη και θα πρέπει ε, να δούμε εκεί μια εξέλιξη ανησυχητική, διότι η, η φωνή των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της κοινωνίας των πολιτών είναι κάτι το ουσιαστικό για την αξία που έχει η ελευθερία έκφρασης. Υποστηρίζω βεβαίως όλα τα, όλους τους συμβιβασμούς, όλα τα συμβιβαστικά κείμενα πάνω στα οποία εργαστήκαμε. Ελπίζω ότι μέχρι τη Δευτέρα δεν θα υπάρξουν αλλαγές στη στάση των άλλων πολιτικών ομάδων. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο σχετικά με το θέμα αυτό και ελπίζω ότι πάνω στα σημεία αυτά θα έχουμε ε, μια συνεκτική ε, ψήφο τη Δευτέρα. Σχετικά με τις άλλες τροπολογίες, έχω μια κατάλογο ψηφοφοριών ε, που ακολουθεί τις αρχές που ενέπνευσαν τη σύνταξη της έκθεσης και τις συμβιβαστικές τροπολογίες που ανέφερα ήδη στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων που είχαμε. Θα υποστηρίξω μόνο τις τροπολογίες που είναι σαφείς ε, συνεκτικές και που φέρνουν κάτι το καινούριο, κάτι το νέο στην έκθεση, που συμπληρώνουν κατά κάποιο τρόπο την έκθεση. Δεν θα υποστηρίξω τις τροπολογίες που αναφέρονται ε, σε τρίτες χώρες και κυρίως αυτές που αναφέρονται σε κράτη-μέλη. Το εξήγησα αυτό στις συναντήσεις μας ότι αυτή η έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι ε, το ίδιο θέμα με το οποίο ασχολείται η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Δεν πρέπει να εκφέρουμε κριτικές στα κράτη-μέλη ανάλογα με τις πολιτικές μας ευαισθήσεις, αν δεν μας αρέσει μια κυβέρνηση που είναι από άλλη χρειά. Δεν, αυτό δεν είναι θέμα ε, της έκθεσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε άλλες πολιτικές μάσχες. Δεν πρέπει να χάσουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τα δικαιώματα στην Επιτροπή μας για να πάρουμε ε, εκδίκηση, αν θέλετε, μεταξύ ε, οικογενειών και ομάδων πολιτικών. Ξέρετε πολύ καλά γιατί περί τίνος πρόκειται. Νομίζω ότι ότι είχαμε με όλα τα μέλη της Επιτροπής ενδιαφέρουσες συζητήσεις και τροπολογίες και ελπίζω ότι τη Δευτέρα θα έχουμε ε, μια ψήφο που θα μας δώσει μια, ένα συνεκτικό κείμενο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κύριε Πρέτα. Θα δώσουμε τον λόγο ε, στους ε, κοιόδης ο κύριος Παλβέρη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Πρέτα για την εξαιρετική δουλειά που έκανε μέχρι τώρα. Και όπως είπε, παρά το μεγάλο αριθμό των τροπολογιών που κατατέθηκαν, μπόρεσε να καταλήξει σε συνένεση των πολιτικών ομάδων μέσω συμβαστικών τροπολογιών. Σε ό,τι αφορά τη δική μου ομάδα, Νομίζω ότι μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι, γιατί ένα μεγάλο μέρο των προτεραιοτήτων μα έχουν συμπεριληφθεί στι συμβαστικέ τροπολογίε. Θα αναφέρω κάποιε. Τη σημασία του να προβλέπουμε μακροπρόθεσμες πολιτικές και να δημιουργούμε ανθρωπιστικού διαδρόμου και για την απελευθέρωση των καθεστώτων θεωρήσεων, το θέμα τη αναγνώριση των δεσμευτικών νομικών μέσων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για τις επιχειρήσεις, η πρόληψη και η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και τη σημασία των διεθνών προτύπων εργασίας για την προστασία των εργαζομένων και τέλος την αναγκαιότητα για τα focal point και τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι ανεξάρτητες και να έχουν άμεσες επαφές με την κοινωνία των πολιτών. Φυσικά παραμένουν ανοιχτά ορισμένα ζητήματα που επίσης είναι προτεραιότητα για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες και δεν έχουν συμπεριληφθεί στους συμβασμούς. Και για όλα αυτά θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή την επόμενη Δευτέρα. Εγώ έχω κατά νου την κάθε καταδίκη ε, της ε, θανατικής ποινής και το σημαντικό θέμα των απαραγωγικών δικαιωμάτων, τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία, των ε, δικαιωμάτων των ΛΟΑΔ και την εφαρμογή των ρήτρας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι θέματα που για μας είναι πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα θα τα δούμε και τη Δευτέρα, όμως ε, εν γέννη είμαστε ικανοποιημένοι με τις συμβαστικές τροπολογίες τις οποίες έχουμε επιτύχει και ευχαριστούμε τον κύριο Πρέντα και όλους τους και για το καλό κλίμα, για την καλή ατμόσφαιρα συνεργασίας και εγώ πιστεύω ότι τη Δευτέρα θα μπορέσουμε να έχουμε μια ψηφοφορία με μεγάλη συνένεση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Προσωπείτε την κυρία Λοχμπίλερ. Γιατί δεν είναι εδώ. Παρακαλώ, κύριε Τέιλορ. Ευχαριστώ. Όπως σωστά παρατηρήσατε, η κυρία Λοχμπίλερ ε, από τους Πράσινους δεν είναι εδώ. Είναι σε μια αντιπροσωπεία ε, στον ε, ΟΑΣΕ και λαμβάνει χώρα ταυτόχρονα. Μου είπε λοιπόν να, πω εκ μέρου τη τα εξή. Καταρχήν ευχαριστεί τον κύριο Πρέντα, τον εισηγητή και του υπόλοιπου σκιώδε για την συνεργασία για την έκθεση. Πολύ σημαντικό για τους πράσινους ήταν μεταξύ άλλων για την έκθεση αυτή του χρονού θέματα όπως το ότι συρρυκνώνε το χώρο για την κοινωνία των πολιτών, η μετανάστευση, τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα καθώς και τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ατιμορρυσία, η εφαρπαγή της γης και η εμπορία ανθρώπων για να αναφέρω Κάποια από αυτά τα θέματα επίσης αντικατοπτρίζονται στις συμβιβαστικές τροπολογίες και κυρίως ό,τι αφορά την ε, υποστήριξη για την ICC ε, και την καταπολέμηση της ατιμορρησίας. Επίσης υπάρχει ο συμβιβασμός ε, για θέματα αθλητισμού και τη σχέση του με τα ανθρώπινα δικαιώματα που θέτει αυτό το θέμα ως απόν από την αρχική έκθεση, από το αρχικό σχέδιο έκθεσης το όλο ένα και πιο δύσκολο περιβάλλον για την κοινωνία των πολιτών σε όλο τον κόσμο επίσης αναγνωρίζεται. Παρ' όλα αυτά, σε κάποια άλλα ζητήματα, όπως η μετανάστευση και η επιχειρήση και τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα θέλαμε πιο ισχυρή διατύπωση. Παραδείγματο χάρη, συμπεριλαμβάνοντας και τις ευρωπαϊκές ευθύνες. Συνάδελφός μου ανυπομονή για την υιοθέτηση αυτή τη εκθέση στην επόμενη συνεδρίαση τη ΑΦΕ τη Δευτέρα και την ψηφοφορία στην Ολομέλεια το Δεκέμβριο. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Thank you very much. Mr. Ευχαριστώ, κύριος Οσεβίτσιου. Thank you, Good morning to everybody. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σε όλους. Θα ήθελα να συγχαρώ τον ε, συνάδελφο Κρίστιαν Πρέντα ε, για την ολοκληρωμένη εξήγηση του εξονόματος του συναδέλφου Μισελ που είναι σκιώδης εισηγητής ενημερώθηκε ότι οι τροπολογίες που συμφωνήθηκαν και είναι 48 νομίζω είναι μια καλή βάση ε, για να έχουμε μια συμφωνία συμβιβαστική. Έχουμε μερικές αμφιβολίες για την τελευταία τροπολογία, την τροπολογία 48, αλλά νομίζω ότι εν ευθέτω χρόνο θα βρούμε την κατάλληλη γλώσσα, την κατάλληλη διατύπωση για τις τελευταίες γραμμές αυτού του συμβιβαστικού κειμένου. Και ελπίζω ότι οι συνάδελφοι θα βρουν μια καλή συμφωνία μεταξύ τους και θα ήθελα άλλη μια φορά να συγχαρώ τον συνάδελφο Πρέντα και ελπίζουμε ότι θα έχουμε το τελικό κείμενο το οποίο θα μπορούμε να υποστηρίξουμε. Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ τον κύριο εισηγητή και τους Σκιώδης για το έργο τους και θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο έχει να κάνει με τη διάρθρωση της εμπορικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την πολιτική της πρόθεσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο η μόνιμη συμπερίληψη ρητρών ε, σε εμπορικέ συμφωνίε που ε, ακριβώ στοχεύουν στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, θα πρέπει να αποτελούν ένα από το καλύτερο τρόπο εγγύηση μια καλύτερη και πιο δίκαιη παγκοσμιοποίηση τη οικονομία. Και αυτή η διάρθρωση μεταξύ εμπορική πολιτική και προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων νομίζω ότι θα πρέπει να λαμβάνει μεγαλύτερη σημασία στο μέλλον. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητά διάφορες εμπορικές ε, συμφωνίες ε, και μέσω του ΠΟΕ αλλά και σε διμερές επίπεδο και επίσης ε, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να θέσει απαιτήσει σε σχέση με την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις περιοχές και με τις χώρες με τις οποίες συνάπτει αυτές τις συμφωνίες. Εγώ νομίζω ότι στο μέλλον θα πρέπει να παγιώσουμε αυτή την οδό, να ακολουθήσουμε αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλετε να απαντήσετε. Ε, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τις ε, προτάσεις τους όσον αφορά τις ε, συμβιβαστικές αυτές προτάσεις. Όσον αφορά τη συμβαστική 48, την τελευταία, και για να είμαι σαφής, εδώ ουσιαστικά πρόκειται για την τελευταία ε, φράση ουσιαστικά αυτής της ε, συμβιβαστικής πρότασης, κυρίως ε, τις τελευταίες λέξεις που αναφέρεται σε μια προσπάθεια να διαλυκανθούν αυτές οι διατυπώσεις και σας διευκρινίζω ότι πρόκειται για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δηλαδή ακριβώς πριν τη φράση αυτή την επίμαχη μιλάμε για τους ε, μηχανισμούς αυτούς τους ε, χρηματοδοτικούς για να καταπολεμήσουμε την διαφθορά. Η διαφθορά βεβαίως είναι ένα πολιτικό θέμα που έχει επιπτώσεις και αντίκτυπο στα δικαιώματα, πρόκειται όμως για ένα πολιτικό θέμα που επηρεάζει τα δικαιώματα. Με αυτήν την προσθήκη απομακρυνόμαστε ακόμα περισσότερο από την ουσία του θέματό μας. Γι' αυτό και πιστεύω ότι αυτή η διατύπωση αρκεί κατά κάποιο τρόπο δείχνει ότι ανησυχούμε. Σε καμία περίπτωση όμως δεν πρέπει να εμποδίσουμε μία συμφωνία για ένα θέμα που αφορά κάτι άλλο. Πρόκειται για ε, φόρους και όχι για δικαιώματα. Εν πάση περιπτώσει. Να δούμε μήπως βρούμε την καταπληκτική αυτή λέξη, η διατύπωση η οποία θα βοηθήσει τους φιλελεύθερους να ξεπεράσουν αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Ίσως το Σαββατοκύριακο να γίνει το θαύμα, να βρεθεί η θαυματουργή αυτή η λέξη που θα βοηθήσει όλους να υπερψηφίσουν αυτή τη συμβαστική πρόταση και να μην περάσουμε σε ελεύθερη ψηφοφορία. Κύριε Πρέδα, είναι μαζί μας και η κυρία Ελίζα τη με συγχωρείτε. Ξέρετε, είναι γραμμένο στα αγγλικά το μικρό σας όνομα. Ζητώ συγγνώμη λοιπόν που πρόφερα λάθος ε, το επιθετό σας. Ε, είναι επικεφαλής ε, του Τμήματος για τις Κατευθυντήριες Γραμμές για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολυμερούς συνεργασίας της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μ' αρέσει όταν μου φωνάζουν τάιζουν. Δεν είμαι ακόμα διευθύντρια, είμαι επικεφαλής ε, αυτού του τμήματος. Α, συγγνώμη, ε, αυτό νόμιζα ότι είπα. Ναι, ναι, είστε υπεύθυνοι επικεφαλής. Α, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε. Για την στρατηγική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ήθελα να πάρω το λόγο για να ευχαριστήσω τον κύριο Πρέντα, να τον συγχαρώ για την ποιότητα της έκθεσής του. Την βρίσκουμε πολύ ευανάγνωστη, τη βρίσκουμε πολύ συγκεκριμένη, αφορά το συγκεκριμένο θέμα και όσον αφορά την επόμενη ετήσια έκθεση θα προσπαθήσουμε ως προς την ουσία να είμαστε λίγο πιο ε, αναλυτικοί όσον αφορά τη γεωγραφική προσέγγιση, να μην είμαστε τόσο περιγραφικοί, να δούμε ποιες είναι οι προκλήσεις, ποιες είναι οι δυσκολίες και να δούμε αν υπάρχουν και κάποιες επιπτώσεις στις δικές μας δραστηριότητες. Θα ακολουθήσουμε επίσης και τις δικές σας συστάσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, να δούμε δηλαδή καλύτερα τα αποτελέσματα, να στοχεύουμε τα αποτελέσματα και να υλοποιήσουμε τις επιπτώσεις της στρατηγικής μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει η Λοιπόν, ολοκληρώνουμε και αυτό το θέμα και θα αναμένουμε την ψηφοφορία στις 16 Νοεμβρίου στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Ευχαριστούμε, κύριε Πρέντα, και με το καλό. Bueno, eh, el Το επόμενο σημείο είναι να σας ενημερώσουμε σχετικά με το ταξίδι μας στη Γενική Συνέλευση των Ενώνων Εθνών την εβδομάδα της 1ης Νοεμβρίου. Πρόκειται για μια κοινή αντιπροσωπεία μεταξύ των Επιτροπών ε, Εξωτερικών Υποθέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων γίνεται ετησίω και μπορέσαμε να συναντηθούμε με, τις, με υψηλούς, υψηλά ειστάμενους στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών. Συναντήσαμε άτομα που είναι υπεύθυνα για τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά συζητήσαμε και προβλήματα που έχουν σχέση με την επίλυση σειράξεων, γεωγραφικές και θεματικές περιοχές, και φυσικά συναντηθήκαμε και με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Μπανκιμούν και τις υπεύθυνε από το UN Women και κάποιους ε, ηθήνοντες για τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης όπως και της Τρίτης Επιτροπής που εντός της Γενικής Συνέλευσης είναι υπεύθυνη για τις χώρες Μαγκρέμπ, για την ασφάλεια στη Βορειοαφρική κτλ. Νομίζω ότι οι συνεδριάσεις ήταν πολύ ψηλού επίπεδου και νομίζω ότι στα Ηνωμένα Έθνη συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο το πόσο σημαντικό είναι ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά το ίδιο ισχύει και από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυξημένη συνειδητοποίηση για το σημαντικό ρόλο που παίζουν τα Ηνωμένα Έθνη παρόλα τα προβλήματα. Ο Γενικό Γραμματέας ήταν σαφέστατος. Ζήτησε μια διαβρεμένη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένων Εθνών και μίλησε ε, για κοινέ προκλήσεις. και για τους οργανισμούς. Μιλήσαμε φυσικά πολύ για το θέμα της Συρίας, για τους πρόσφυγες, που βέβαια βάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση σε, σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση ενώπιον του υπόλοιπου κόσμου. Έχουμε χάσει πάρα πολύ την αξιοπιστή μας. ήταν πολύ πλοκό το θέμα τη αξιοπιστία τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολλού τομεί. Για τα ανθρώπινα δικαιώματα διατηρούσαμε ένα επίπεδο και εγώ νομίζω ότι με την κρίση των προσφύγων ε, μα έκανε να χάσουμε πάρα πολλού πόντου στο ότι δεν χειριστήκαμε κατάλληλα την κρίση των προσφύγων δηλαδή. Υπάρχουν πολλά προβλήματα προπολογισμού στους οργανισμούς και όλο ένα και περισσότερα προβλήματα. Έχουμε και λιγότερους πόρους. Και βέβαια και οι λίγοι πόροι που υπάρχουν ε, δεν φτάνουν τη στιγμή που πρέπει. Έχουμε λοιπόν περισσότερα προβλήματα, λιγότερους πόρους και καθυστερούν και οι πόροι. Είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη λοιπόν η κατάσταση και όλοι ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει μια μεγαλύτερη προσπάθεια. Πρόεδρος της ε, Γενικής Συνέλευσης, ο κ. Λικέτοφ, τον οποίο είχαμε ένα μακροσκελές γεύμα, προσέγγισε έντονα τα θέματα της ε, κλιματικής αλλαγής και είπε ότι μάλλον είναι η τελευταία ευκαιρία μας να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι πραγματικά χρήσιμο για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και ότι το Παρίσι είναι μια στιγμή κλειδί για το ζήτημα αυτό. Τώρα, όσοι ενδιαφερόμαστε περισσότερο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, είχαμε μια πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα που λέγεται Human Rights Up Front. Ο στόχος είναι να τεθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στο υψηλότερο επίπεδο ανάλυσης, έτσι ώστε τα Ηνωμένα Έθνη να παρεμβαίνουν πριν να έχει ξεσπάσει η καταστροφή. Δηλαδή να υπάρχει ένα μόνιμο σύστημα ανάλυσης ε, και τα ανθρώπινα δικαιώματα να είναι σε θερμόμετρο που μετρούν σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι διάφορες κοινωνίες ή διάφορες σειράξεις, έτσι ώστε να μπορούμε να παρεμβαίνουμε πριν να έχει ξεσπάσει η καταστροφή. Και αυτό το είχαμε κάνει στη Συρία όταν έπρεπε, μάλλον δεν είχαμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση και ούτε στη Λιβύη και το ίδιο και για την Ιεμένη αλλά καθώς δεν το κάναμε αυτό, τελικά οι σειράξει μεγενθύνονται και όταν ξεσπούν είναι πολύ πιο δύσκολο να τις αντιμετωπίσουμε. Έτσι λοιπόν αυτή η πρωτοβουλία στην οποία εργάζονται άνθρωποι από το γραφείο του Μπανκιμού να έχει αυτό το στόχο. Και θέλει να θέσει τον πυλώνα ανθρώπινα δικαιώματα σε ίδιο επίπεδο με τον πυλώνα της ειρήνης, της ασφάλειας και της ανάπτυξης. Αυτοί οι τέσσερις πυλώνες δηλαδή να έχουν την ίδια σημασία και ισχύ. Φυσικά όλο αυτό έχει να κάνει και με τη μεταρρύθμιση του Γενικού Συστήματος των ΗΕ. Εθνών και υπάρχουν διάφορες συζητήσεις. Κάποιοι από το, ε, τους ανθρώπους με τους οποίους συναντηθήκαμε έδειξαν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το δικό μας έργο και τους καλέσαμε να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις μας σε διάφορες χρονικές στιγμές και Νομίζω ότι συντονισμένη δουλειά με τα Ηνωμένα Έθνη θα είναι κάτι πολύ θετικό και για μας, για το δικό μας έργο. Υπάρχουν πάρα πολλά άλλα πράγματα που θα μπορούσα να σας αναφέρω, αλλά καθώς ε, είναι εδώ τουλάχιστον ο κ. Στελίτσιος που με συνόδευσε στην αποστολή, θα του δώσω το λόγο για να δώσει και αυτός από την πλευρά του κάποιες εξηγήσεις. Σας ευχαριστώ κ. your... Ευχαριστώ. Βεβαίως με την αξιολόγηση σας συμφωνώ σχετικά με την επίσκεψή μας στα Ηνωμένα Έθνη. Αυτή είναι νομίζω μεγάλη ευκαιρία να πάει κανείς στα Ηνωμένα Έθνη για να δει όλα τα παγκόσμια θέματα συνδεδεμένα ταυτόχρονα ε, και όλες τις χώρες και όλες οι απόψεις που αντιπροσωπεύονται ε, από από σημειώσεις που πήρα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ορισμένες φορές υποτιμούμε την σημασία και την χρησιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα παγκόσμια θέματα. Εκτιμηθήκαμε ως οργάνωση, ως θεσμό, θεσμικό όργανο πάρα πολύ και οι αξιωματούχοι τους οποίους συναντήσαμε όχι μόνο μία φορά αλλά πάρα πολλές φορές επανέλαβαν την εκτίμησή τους και την ε, σημασία, το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα παγκόσμια θέματα των Ηνωμένων Εθνών για την ενημέρωσή σας Έχουμε για την ώρα τέσσερα μέλη, τέσσερα κράτη-μέλη που αντιπροσωπεύονται στο Συμβούλιο Ασφαλείας και στο προσεχές μέλλον θα έχουμε τρία και σε άλλο στάδιο πέντε, σε απότερο στάδιο. Για να μην αναφέρω ε, τις εκλογές, τις επερχόμενες εκλογές για το Γενικό Γραμματέα που υπάρχει μια γραπτή συμφωνία ότι η θέση αυτή ανήκει μάλλον ε, σε ανατολικό ευρωπαϊκά κράτη και περιμένουμε αυτήν την άσκηση, αυτό το εγχείρημα το ενδιαφέρον ε, σύντομα. Ξέρετε ότι υπάρχει ένας μεγάλος κατάλογος υποψηφίων που μπορούμε εμείς οι ίδιοι να αξιολογήσουμε. Θα είναι μια, μια ενδιαφέρουσα στιγμή για όλους μας. Σύμφωνο μαζί σας ότι πρέπει και εμείς να συνεχίσουμε να καλούμε στις συνεδριάσεις μας στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο αυτούς τους υψηλούς αξιωματούχους από τα Ηνωμένα Έθνη για να φέρω παραμπτός χάρη τον πρέσβη του Μαρόκου που συναντήσαμε και που είναι επικεφαλής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών και νομίζω ότι θα μπορούσαμε έτσι να ανταλλάξουμε απόψεις, μπορούσαμε να οργανώσουμε ε, νομίζω μια ειδική εκδήλωση για να εστιαστούμε στις ε, δραστηριότητες της σχετικές των Ηνωμένων Εθνών. Θα πρέπει λοιπόν να ε, πηγαίνουμε και να τους συναντούμε και να τους καλούμε εδώ, διότι αυτό είναι προστιθέμενη αξία. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια προσωπική επαφή και να ανταλλάσσουμε απόψεις προφορικά και όχι με γραπτές σημειώσεις σε διαφορετικές περιστάσεις ε, και νομίζω ότι ερχόμενοι εδώ θα αλλάξει η κατάσταση. Νομίζω ότι η ομάδα ήταν πάρα πολύ ικανοποιητική, το ταξίδι πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πολύ. Αν δεν υπάρχουν ερωτήσεις, από ό,τι φαίνεται όχι, θα κάνουμε 10 λεπτά διάλειμμα. Πριν να ξεκινήσουμε με το επόμενο σημείο, ήδη έχει φτάσει προς και κλειμένος ο κύριο Βασίρ και η κυρία Ρόγολ. Θα ήθελα ένα λεπτό να τοποθετηθούν για το προηγούμενο σημείο δήλωση για το ταξίδι μας στη Νέα Υόρκη, στη Γενική Συνέλευση των Εθνών. Έχετε ένα λεπτό, κύριε Βασίλου. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, θα ήθελα πραγματικά να συγχαρώ την εργασία όλων αυτών ε, των μελών του προσωπικού, των συνεργατών μας εδώ και εδώ και στην Νέα Υόρκη την προετοιμασία αυτής της αποστολής. Ήταν εξαιρετικά σημαντική και εξαιρετικά επιτυχής στενή συνεργασία για την οποία υπογραμμίσατε το πόσο σημαντική είναι μεταξύ ημών και των Ηνωμένων Εθνών γιατί έχουμε κοινά θέματα και τους πρόσφυγες, ε, ισότητα των φύλων, την ειρήνη, την ασφάλεια, την αναπτυξιακή βοήθεια. Η ομάδα μου παρόλα αυτά υποστηρίζει και την μεταρρύθμιση των Ηνωμένων Εθνών έτσι ώστε να υπάρξει περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη αποτελεσματικότητα για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις μεγάλες προκλήσεις, τις παγκόσμιες. Γενικός Γραμματέας, ο οποίος ε, θα εκλεγεί το 2016, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να επιλεγεί ο πιο κατάλληλος, ο πιο αρμόδιος, άσχετα από το που προέρχεται. Το θέμα των παγωμένων σειράξεων, οι οποίες από τη φύση τους ε, δεν έχουν επιληθεί εδώ και πολύ ε, μεγάλο χρονικό διάστημα και μάλιστα αποκρισταλώνουν πολύ σημαντικές εντάσεις και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δει πώς μπορεί να συνεισφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη μεταρρύθμιση των Ηνωμένων Εθνών χωρίς βεβαίως να υπονομεύσει εδώ τα δικαιώματα των μεμονωμένων κρατών μελών διότι βεβαίως μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα αυτό των ΗΠΑ μόνο με ομοφωνία. Και σαφώς είναι καθοριστικό για την κυρίαρχη εξωτερική πολιτική του κάθε κράτους να συγκεράσει αυτό το κοινό συμφέρον με τα εθνικά του συμφέροντα. Γι' αυτό και ο ενισχυμένος ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εσωτερικό των Ηνωμένων Εθνών είναι πολύ σημαντικό, όπως και το θέμα της ε, μίας έδρας στο Συμβούλιο Ασφαλείας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο θα διασφαλίσει ότι τα Ηνωμένα Έθνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη αλλά και άλλοι διεθνείς οργανισμοί θα μπορέσουν να συνεργαστούν με τον καλύτερο τρόπο για την επίλυση των μεγάλων προβλημάτων. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα είμαι πολύ σύντομη, γιατί βεβαίως ε, ήταν μια πάρα πολύ επιτυχής ε, αποστολή. Θα κάνω δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, δεν είναι δική μας αρμοδιότητα βεβαίως, αλλά όλες οι ανταλλαγές ε, επαφές που είχαμε μας έδειξαν ότι είναι πάρα πολύ επίγουσα η μεταρρύθμιση των Ηνωμένων Εθνών. Η δική μας εμπειρία από συνεργασία εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση μας δείχνουν ότι μπορούμε να συνεργαστούμε καλύτερα με ένα μεταρρυθμισμένο οργανισμό. Δεύτερον, και εγώ με όλες αυτές τις επαφές που είχαμε συνειδητοποίησα ότι αυτά που συμβαίνουν σήμερα με τους πρόσφυγες στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίοι βεβαίως ε, προσπαθούν να ξεφύγουν από σημαντικές κρίσεις αλλού στον κόσμο, να αποφύγουν δύσκολες καταστάσεις, μας οδηγούν στη διαπίστωση ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο προληπτικοί. Εμείς εδώ, στην Επιτροπή μας, σαφώς και θα πρέπει να είμαστε πιο προληπτικοί, γιατί τα ανθρώπινα δικαιώματα και η προστασία τους έχουν μεγάλη συνάρτηση με την πρόβλεψη τέτοιων καταστάσεων. Καταλαβαίνετε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα αυτών που προσπαθούν να διαφύγουν από πόλεμο και από τέτοιες ακραίες βίες καταστάσεις προστατεύονται πολύ καλύτερα εάν δεν είχαν βρεθεί σε αυτή την κατάσταση. Σήμερα λοιπόν βλέπουμε ότι αν ήμασταν πιο προληπτικοί θα είχαμε πολύ λιγότερο πρόβλημα να αντιμετωπίσουμε. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Η αλήθεια είναι ότι αφού επισκεφθήκαμε τα Ηνωμένα Έθνη, και υποθέτω ότι θα με καταλάβει πλήρω ε, και η κυρία δικαστή. Μετά λοιπόν την επίσκεψη στα Ηνωμένα Έθνη, παρόλε τι ε, κριτικέ, με τι οποίε μπορούμε να συμφωνήσουμε ή όχι, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι αν δεν υπήρχαν θα έπρεπε να φεύγουμε τουλάχιστον. Ευτυχώ ε, που συνεχίσουμε να έχουμε τα Ηνωμένα Έθνη. Τώρα λοιπόν περνάμε σε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για την Επιτροπή μας. Έχουμε μαζί μας ε, την κυρία Μέρι Ντέιβις. Της ανέθεσαν τα Ηνωμένα Έθνη να κάνει μία έρευνα για τη σύραξη στη Γάζα από τις 7 ε, Ιουνίου μέχρι ε, τον Αύγουστο του 2014 μέχρι τις 26 Αυγούστου έχει παρουσιάσει τον Ιούνιο του 2015 την έκθεσή της στα Ηνωμένα Έθνη και ξέρετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Σεπτέμβριο του 2014 καταδίκασε σφοδρά τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της σύραξης και ένα δεύτερο ψήφισμα το Σεπτέμβριο του 2015 ζήτησε επίμονα από την ύπατη ε, εκπρόσωπο να αναλάβει δράση και να εφαρμόσει τις συστάσεις που διατυπώθηκαν τόσο από τη δική σας έκθεση όσο και βάσει των αποφάσεων αυτού του Κοινοβουλίου. Για μας είναι κεφαλαιόδου σημασία να δούμε ποια είναι η άποψή σας από πρώτο χέρι και σας ευχαριστούμε που ήρθατε μέχρι εδώ για να μας κοινοποιήσετε τα όσα μπορέσατε να διαπιστώσετε. Σας ευχαριστώ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι, καλημέρα σα. Λέγομαι Μέρη Μακαλαντήρη, είμαι πρόεδρο τη Ανεξάρτητη Εξεταστική Επιτροπή του ΙΕ για τη σύραξη στη Γάζα του 2014. Με τιμά η πρόσκληση να απευθυνθώ σε εσά σήμερα το πρωί για την έκθεση της Εξεταστική επιτροπή που εκδόθηκε τον προηγούμενο Ιόνιο. Θα σας ε, μιλήσω για το έργο της Επιτροπής και θα αναφέρω τα κύρια πορίσματα και τις συστάσεις και κατόπιν κατανοώ ότι κατόπιν θα υπάρχει μια ανταλλαγή απόψεων ε, σε σχέση με τα συμπεράσματα για την παραβίαση του ανθρωπιστικού δικαίου και την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κάτι που μπορεί να έχει γίνει και από τους Ισραηλινούς αλλά και από τις Παλαιστινικές ομάδες κατά το καλοκαίρι του 2014. Ξέρω ότι η άνοδος ε, της βίας ε, τις τελευταίες ε, εβδομάδες είναι πολύ ανησυχητική. Επομένως, εμένα με οδηγεί στο να αναφερθώ στο ότι είναι πήγον να δράσουμε τώρα για να σταματήσουμε την αιματοχυσία. Τι η Εξεταστική Επιτροπή τι δεν ήταν. Ε, ο Δ. και εγώ δεν ε, προσπαθήσαμε να έχουμε μια ετοιμιγορία ενοχής, να αποδέσουμε μια ετοιμιγορία ενοχής για τα, κάποια από τα μέρη. Δεν ε, ήταν μια δικαστική διαδικασία, δεν υπήρχαν μαρτυρίες, αλλά βασιστήκαμε σε πληροφορίες που μας δόθηκαν στην έκθεση δεν μιλάμε για αποδεικτικά στοιχεία. Αυτό που συλλέξαμε αντίθετα και με ένα πολύ σχολαστικό τρόπο έχει να κάνει με υλικό που μπορούν να μας δείξουν τον τρόπο για μια ευρύτερη έρευνα για το τι έγινε το καλοκαίρι του 2014 στη Γάζα, στη Δυτική Όχθη και στην Ιερουσαλήμ και στο Ισραήλ για να καθορίσουμε αν κάποια συμπεριφορά από τις ε, δύο πλευρές ε, παραβίασε το δίκαιο. Εγώ ε, δεν νιώθω άνετα ουσιαστικά να λέω πράγματα πέρα από αυτά που λέγονται στην έκθεση και ξέρω και ότι ο συνάδελφός μου νιώθει το ίδιο. Εμείς στο κείμενο έχουμε ακολουθήσει πολύ προσεκτική διατύπωση αλλά θα προσπαθήσω να σας τονίσω κάποια σημεία τώρα και θέλω να απογραμμίσω ότι η σύντομη έκθεση συνοδεύεται από ένα παράρτημα 103 σελίδων όπου αναφερόνται λεπτομερώς πολλά συγκεκριμένα περιστατικά που εξετάσαμε και η ουσία των μαρτυριών των μαρτύρων και ουσιαστικά γίνεται και μία αξιολόγηση. Εργαστήκαμε πάρα πολύ σκληρά για πολλούς μήνες ε, σε αυτή την Επιτροπή γιατί πιστεύουμε ότι τα θύματα και από τις δύο πλευρές πρέπει να ακουστούν. Είναι πηγή ε, ανησυχία και λύπης που δεν μπορέσαμε να ταξιδέψουμε στο Ισραήλ και στα κατεχόμενα παλαιστινικά εδάφη για να τους συναντήσουμε από κοντά. Αλλά αυτό ε, απλώς ε, μας όπλησε με ισχυρότερη βούληση για να δώσουμε ε, στα θύματα ένα φόρουμ, ένα βήμα όπου θα μπορούσαν να ακουστούν οι ιστορίες τους. Ακούσαμε μαρτυρίες από πολλούς ανθρώπους που θέλουν ο κόσμος να αναγνωρίσει τα δεινά τους και θέλουν να έρθουν στα Ηνωμένα Έθνη για να καταθέσουν τη μαρτυρία τους προκειμένου να αναζητήσουν δικαιοσύνη και ειρήνη. Επίσης, ε, νομίζω ότι ε, τον Ιούλιο του 2014 ο πατέρας ε, που ξύπνησε στο νοσοκομείο και έμαθε τα παιδιά του και αδελφοί του και μητέρα του είχαν όλοι πεθάνει. Συνολικά 19 άτομα της οικογένειάς του, 19 μέλη της οικογένειάς του και είπε ακόμη και αυτοί που επιβιώσαμε πεθάναμε εκείνη την ημέρα και νομίζω ότι ε, νεαρός άνθρωπος στην Γάζα, ε, το οποίο εκτέλεσε τον πατέρα γιατί θεωρεί το συνεργάτης και ε, ανέφερε ότι δεν είχε καμία προοπτική στη ζωή. Η αρβωνιαστικιά του είχε ακυρώσει το γάμο και είχε χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες να βρει εργασία. Η ζωή έχει γίνει αδύνατη για την οικογένειά μου λόγω του στιγματισμού από την κοινωνία και ζήτησε από τους επιτρόπους να πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να αυτοκτονήσει και πιστεύω ότι μία, και, έχω, και σκέφτομαι μάλλον, μία Σιλενή μητέρα, ε, το παιδί της 4 χρονών σκοτώθηκε από χτύπημα ενώ έπαιζε στο σπίτι του. Οι άνθρωποι που ζουν στο Ισραήλ θέλουμε να ζούμε ειρηνικά και όχι από την απειλή τη τρομοκρατία, μα είπε. Θέλω οι γείτονέ μα στη Γάζα να έχουν μια καλή και ευτυχισμένη ζωή και τα παιδιά του να πάνε στο σχολείο. Τώρα, νομίζω ότι αυτό το οποίο μπορούμε να ελπίζουμε από όλη αυτή τη μακρά διαδικασία της εξέτασης είναι ότι κάπως ε, προχωρήσαμε λίγο περισσότερο ε, στον τομέα της δικαιοσύνης και της ειρήνης, κυρίως καλώντας ε, τις κυβερνήσεις όπως της Ευρωπαϊκής Ένωσης από κοινού να καλέσουν για αλλαγή των πολιτικών σε σχέση με την χρήση των εκρηκτικών όπλων, κυρίως σε κατοικημένες περιοχές όπως τη Γάζα και να λογοδοτήσουν ε, όσοι δεν προστατεύουν ε, τις ε, ζωές των αμάχων. Κυρίως είδαμε τι συνέβη στη Γάζα και στο Ισραήλ τον Ιούλιο του 2014. Θα αναφέρω και κάποια άλλα στοιχεία που μας ενσύχησαν στη σύραξη του 2014. Καταρχήν, ε, τεράστια αύξηση στη χρήση των ε, πυροβόλων όπλων ε, και η καταστροφή οικογενειών και σπιτιών. Είχαμε πολλές οικογένειες, όλα τα μέλη τους ξεκληρίστηκαν όταν έπεσαν βόμβες στο σπίτι τους ενώ γιορτάζαν το Ραμαζάνι. Αυτές οι επιθέσεις είχαν μεγάλες συνέπειες για τα παιδιά. Περίπου 551 παιδιά ε, κατέληξαν στη Γάζα τότε. Καταστράφηκαν πάρα πολλές ε, κατοικίες ε, και ε, στοχεύτηκαν ε, σπίτια που ανήκαν σε πολιτικούς. Έτσι λοιπόν ε, αυτό μας δείχνει ότι υπήρχαν κάποιοι στρατιωτικοί στόχοι που όμως ήταν πιο επεκτατικοί από ό,τι προβλέπεται στο διεθνές δίκαιο και τη στιγμή των επιθέσεων όταν ήταν πιθανό να είναι στο σπίτι οικογένειας τους η χρήση τεραστίων βομβών σε πυκνοκατοικημένες περιοχές με το συνδυασμό ότι αυτέ οι θανατηφόρες επιθέσεις συνεχίστηκαν για εβδομάδες ενώ είχαν ε, άμεσο αντίκτυπο στους αμάχου και αυτό φάνηκε από τις πρώτες ημέρες της σύρεξη. Ε, όλο αυτό ε, μάλλον το, τη θεωρείται ότι μπορεί να ήταν μια ευρύτερη πολιτική ε, και ουσιαστικά οι αποφάσεις ε, λήφθησαν από ξεμετούχους σε ανώτατα κλιμάκια τη κυβέρνησης. Επίσης, ε, είχαμε τεράστιες απώλειες στη Ράφα και σε άλλες πόλεις και ουσιαστικά χρησιμοποιώντας μετρελαιοβόλια όπλα και μπουλντόζες ισοπεδώθηκαν ολόκληρες γειτονιές. Αυτές οι περιοχές ισοπεδώθηκαν η μία μετά την άλλη και αυτό θα να ανησυχία ότι δεν χρειαζόταν από, ε, για στρατιωτικούς λόγους τέτοιες ευρείες ε, καταστροφές ε, στην Ράφα όταν φοβήθηκαν οι Ισραηλινοί ότι είχε συλληφθεί ένας στρατιώτης ε, ουσιαστικά τότε ε, μηδραλιοβόλησαν ολόκληρη την πόλη για ώρες και ε, μπορεί τότε ο Ισραηλινός στρατός να μην σεβάστηκε θεμελιώδεις αρχές του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου. Το 2014 οι ένοπλες ομάδες ε, της Παλαιστίνης έστειλαν μια σειρά πυράβλων ε, στο Ισραήλ. Η μεγάλη πλειοψηφία αυτών των βλημάτων ήταν ρουκέτες χωρίς συστήματα κατεύθυνσης και ουσιαστικά ε, στα εστάλησαν σε πυκνά κατοικημένες περιοχές, ρίχθησαν σε πυκνά κατοικημένες περιοχές του Ισραήλ και θεωρούνταν ε, επιθέσεις χωρίς στόχο. Ε, κάτι ακόμα είχαμε ότι οι Παλαιστίνοι χρησιμοποίησαν ε, ε, ουσιαστικά κάποια τούνελ. Η ανακάλυψη αυτών των τούνελ και η χρήση τους από ένα ομαδες των Παλαιστινίων κατά τη διάρκεια των εχθροψιών δημιούργησε μεγάλο άγχος στους ε, Ισραηλινούς ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να επιτεθούν σε αμάχους. Και μας είπε ένας μάρτυρας ότι όταν υπάρχει ησυχία φοβόμαστε περισσότερο γιατί δεν, μπορούμε, δεν ξέρουμε τι θα βγει από το έδαφος. Επίσης ε, η χρήση ε, των πυρομαχικών από τον Ισραηλινό στρατό στη Δυτική Όχθη οδήγησε σε μεγάλο αριθμό θυμάτων και τραυματιών το 2014. Η έκθεσή μας συστήνει Ισραηλινές ε, αρχές να αναθεωρήσουν τις πολιτικές τους σε σχέση με αυτά τα ε, ζωντανά πυρομαχικά σε κατοικημένες περιοχές. Δυστυχώς οι αρχές ανακοίνωσαν τις τελευταίες εβδομάδες ότι ουσιαστικά χαλαρώνουν αυτούς τους περιορισμούς επειδή ε, έχουμε την εμφάνιση μεγαλύτερης αναταραχής στα κατεχόμενα εδάφη και στην Ιερουσαλήμ. Επίσης η Επιτροπή αναφέρθηκε στο ότι όλα τα μέρη δεν κατόρθωσαν να πετύχουν τη δικαιοσύνη με ένα αποτελεσματικό και διαφανή τρόπο ουσιαστικά δεν χρησιμοποιήθηκαν οι κατάλληλοι μηχανισμοί λογοδοσίας. Όπως είπε ένας ε, Παλαιστίνιος, καθημερινά δολοφονείται η δικαιοσύνη, πεθαίνουμε αργά. Πράγματι, η περίπτωση των τεσσάρων αγοριών που σκοτώθηκαν στην ε, παραλία ε, τόνισε ε, τα πενιχρά αποτελέσματα της δικαστικής έρευνας και δείχνει ότι υπάρχει ανάγκη να υπάρχουν αποτελεσματικοί μηχανισμοί λογοδοσίας σε όλες τις πλευρές. Κατανοούμε ότι πάρα πολλοί μάρτυρες και κάποιοι Παλαιστίνοι που παρευρίσκονταν, αλλά και διεθνείς δημοσιογράφοι που ήταν παρόντες στα σύνορα, ούτε καν έδωσαν καταθέσεις και δεν δημοσιεύθηκαν καν οι συνθήκες ε, και οι εικόνες που δημοσιεύθηκαν παρουσίασαν τα αγόρια ε, ως μαχητές. Έτσι λοιπόν πρέπει να γίνονται αξιοποι... έρευνες που να καταπολεμούν την ατιμορρησία. Ο Dr. Τζένιν και εγώ δράξαμε κάθε δυνατή ευκαιρία για να ευχαριστήσουμε όσους συνεργάστηκαν μαζί μας στην έρευνα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί διέτρεξαν και πολλούς κινδύνους μάλιστα ένας ε, Ισραηλινός, ο Διακόνη, είχε χάσει και τα δύο του πόδια σε μια επίθεση με τριαλιοβόλου στο τέλη του και μάλιστα ταξίδευσε στη Γενέβη για να μας πει την ιστορία του. Φυσικά όσοι κατοικούν στη Γάζα δεν είχαν τέτοια ευκαιρία. Ε, Πάρα πολλοί μάρτυρες ε, είχαν έφεραν ψυχικά τραύματα και Κυρίως έχω κατά νου τον άνθρωπο ο οποίος έχασε από το παιδιά του και την σύζυγό του και τη μητέρα του σε πλήγμα στο σπίτι τους. Τι μπορεί να πει κανείς τον άνθρωπο αυτό όταν υποφέρει τόσο. Αυτοί οι μάρτυρες με τους οποίους συνομιλήσαμε στη Γάζα προσπαθούσαν ε, ουσιαστικά να αντιμετωπίσουν τις ε, συνέπειες ε, της σύραξης. Κάποιος μας είπε, σε βλέπεις αυτό Πεπόνι» Ε, εγώ δεν έχω νερό στο σπίτι μου. Ακούσαμε τραγωδίες και αποθήματα και από τις δύο πλευρές και εγώ πιστεύω ότι παρόλο το μίσος υπήρξαν πάρα πολλοί άνθρωποι που εξέφρασαν συμπάθεια για τους ανθρώπους από την άλλη πλευρά. Μια σημερινή γυναίκα μας είπε ότι θα ήθελε να έχει πιο φιλικές σχέσεις με τους γείτονές του σε αυτή την αδύνατη τρελή κατάσταση. Και μια άλλη σημερινή γυναίκα ήθελε να πει στους ηγέτες και των δύο πλευρών θέλουμε αξιοπρέπεια και ελευθερία αλλά και για την άλλη πλευρά και μια Παλαιστίνια ε, που θρηνούσε το θάνατο του Μοχάμετ Καντήρ, ε, ο οποίος ε, απήχθηκε κάκια ζωντανό στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, είπε «Είμαι μεταξύ των εκατοντάδων γυναικών που έχασαν τα παιδιά τους, έχασα το γιο μου το Μοχάμετ και δεν θα έρθει πίσω από το σχολείο να μου τραγουδήσει. Δεν θέλω καμία άλλη μητέρα να περάσει αυτό που πέρασα εγώ». Και γι' αυτό σας ζητώ να σταθείτε μαζί μας και να έχετε κατά νου όλες τις μητέρες που υποφέρουν. Και ένας Παλαιστινίος γιατρός από τη Γάζα μας είπε ότι ο αδελφός του σκοτώθηκε μαζί με άλλους τρεις ασθενείς όταν ε, έγινε επίθεση στην κλινική. Μας είπε ότι θέλει να υπάρχει ένα πνεύμα συνεργασίας και αδελφοσύνης. Θα διαβάσετε την έκθεση και θα ακούσετε πάρα πολλές φωνές τέτοιων ανθρώπων που θέλουν οι ηγέτες να διαπραγματευτούν μια ασφαλή και μακρόχρονη ειρήνη. Και φυσικά θα πρέπει να θυμόμαστε ότι τα θύματα δεν είναι απλώς νούμερα και παράπλευρες απώλειες, είναι άνθρωποι ξεχωριστοί με ανθρώπινα δικαιώματα και δικαιούνται ε, να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για όλες τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Επιτροπή καλωσορίζει το ψήφισμα που υθετήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου του 2015, κυρίως στον παράγραφο 18, που Ρωτή την είπατε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εργαστεί για την πλήρη εφαρμογή των συστάσεων της έκθεσής μας και καλούμε τη διεθνή κοινότητα και ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση ιδίω να επιταχύνει και να τοικοποιήσει τις προσπάθειες προκειμένου να έχουμε πρότυπα πολιτικής που θα περιορίσουν τη χρήση εκρηκτικών όπλων σε πυκνοκατοικημένες περιοχές προκειμένου να προστατευτούν οι άμαχοι κατά τη διάρκεια των χρυσιών. Επίσης, να υποστηρίξει την, ε, το έργο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου σε σχέση με ε, τα παλαιστινικά κατοικόμενα εδάφη, να ασκήσει διεθνή δικαιοδοσία, να δικάσει τα εγκλήματα σε διεθνή δικαστήρια και να στείλει τους υπόπτους ε, σε ε, Χώρε όπου θα υπάρχει δίκαιη δίκη. Επίσης να προωθήσει το σεβασμό τη υποχρεώσεω των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να σεβαστεί να διασφαλίσει το σεβασμό του Διεθνού ανθρωπιστικού δικαίου στα κατεχόμενα παλαιστινικά εδάφη και στο Ισραήλ σύμφωνα με το άρθρο 1 που υπάρχει στις συνθήκες της Γενέβης. Και θέλω να επιστήσω την προσοχή σου σε μια παρατήρηση του Μπαν Κιμούν του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ την περισσότερη εβδομάδα όταν συναντήθηκε με τον Πίτερ Μάουερ τον πρόεδρο του Διεθνού Σύνθρου Σταυρού, ο Γενικός Γραμματέας, τόνισε ότι το διεθνές δίκαιο σήμερα καταπατείται σε παγκόσμια κλίμακα και ότι η διεθνής κοινότητα αποτυγχάνει να οδηγήσει στη δικαιοσύνη ε, τους εγκληματίες. 60 εκατομμύρια άνθρωπα δεν έχουν στέγη και υπάρχει τεράστια ανάγκη για ανθρωπιστική βοήθεια και δεν φαίνεται ότι η ειρήνη θα έλθει στη Συρία, στο Ισραήλ Ισραήλ στην Ιεμένη και εγώ θα προσθέτω και στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν. Κάλεσε τα κράτη να σταματήσουν τη χρήση βαρέοπλισμού σε κατοικημένες περιοχές. Ο Γενικός Γραμματέας παρατήρησε το εξής. Αυτές ε, οι παραβιάσεις έχουν γίνει τέτοια ρουτίνα και υπάρχει κίνδυνος να πιστέψουν οι άνθρωποι ότι σκόμβος βορβαδισμός των αμάχων και η στόχευση των εργαζομένων στον τομέα της υγείας και ε, ότι στοχεύονται σχολεία και νοσοκομεία είναι αναπόφευκτο αποτέλεσμα της σύραξης. Φτάνει πια, ακόμη και ο πόλεμος έχει κανόνες και ήρθε η ώρα να του εφαρμόσουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμη κυρία Ντέιβις για την περιγραφή την πολύ ζωντανή που μας κάνατε. Έχουμε εδώ μαζί μας τον Αντιπρόεδρο της Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με την Παλαιστίνη, τον κύριο Σιλικιώτη και θα ήθελα να του ζητήσω να πάρει το λόγο. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας. Επίσης έχουμε καλέσει και την ε, αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με το Ισραήλ, όμως ε, δεν βρίσκεται εδώ κάποιος συνάδελφος, μέλος της Επιτροπής εκείνη και έχουμε και προσώπους και από τις δύο πρεσβείες και κατόπιν των ερωτήσεων των βουλευτών θα τους δώσω το λόγο, αλλά τώρα έχουμε το, δίνουμε το λόγο στον αντιπρόεδρο της ε, αντιπροσωπείας με τη σχέση με την Παλαιστίνη. Παρακαλώ. Έλενα, ε, πω καταρχήν ότι δεν είμαι αντιπρόεδρος, είμαι μέλος της delegation, δεν υπήρχε αντιπρόσωπος να είναι παρόν. Εμείς στην ε, ε, συνεδρία της ε, αντιπροσωπείας στο σχέσιο με την Παλαιστίνη έχουμε συζητήσει την έκθεση της κυρία Ντέβης. Πρέπει να την ευχαριστήσουμε πρώτα γιατί αποτυπώνει με πάρα πολύ ξεκάθαρο τρόπο όλες αυτές τις παραβιάσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της επέμβασης στη Γάζα ε, και να πω ότι, να σας θυμίσω ότι είχαμε εγκρίνει και ε, το 2014 έκθεση από το Ευρωκοινοβούλιο όπου είχαμε καταδικάσει αυτές τις παραβιάσεις. Βέβαια είναι σαφής η τελευταία απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου το Σεπτέμβριο του 2015 που ακριβώς καλεί την είπα την εκπρόσωπο να αναλάβει δράση. Ε, ε, εμείς ως αντιπροσωπεία η οποία πρέπει να πω ότι δοκιμάσαμε να, τον περασμένο Μάρτιο να επισκεφτούμε τη Γάζα. Δυστυχώ είναι κάτι που και αυτόν το καταγγείλαμε και στο Ευρωκοινοβούλιο και δημόσια. Ε, δεν μα επιτράπηκε η είσοδο τη αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη σχέση με την Παλαιστίνη να επισκεφτούμε τη Γάζα. Για να δούμε δηλαδή, να έχουμε επαφή με του ανθρώπου, να δούμε από πρώτο χέρι όλα αυτά που ε, <clears throat> συνέβηκαν και συμβαίνουν εκεί είναι ξεκάθαρο ότι είχαμε να κάνουμε με μαζικέ παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εγώ θα έλεγα και κάτι, ανεξάρτητα καμιά φορά μιλούμε για την τρομοκρατία, η οποία είναι καταδικαστία από όλου, ε, πόσο μάλλον όταν εδώ ε, ασκείται μια, ασκήθηκε μια και συνεχίζει να ασκείται στα, στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη μια κρατική τρομοκρατία, διότι δηλαδή, περί αυτού πρόκειται. Όταν μιλούμε για επέμβαση στη Γάζα και αυτά που χρησιμοποίησε ο Ισραηλινό στρατό, μιλούμε για μια ανεπίσημη πλέον κρατική τρομοκρατία, η οποία επέφερε ε, τόσο πολλά θύματα, η οποία δυστυχώ αυτή η βία συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Ε, Εμεί θεωρούμε ότι είπα διεκπρόσωπο για τι εξωτερικέ σχέσει ε, και πρέπει να λάβει δράση, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, πρέπει να πάρει μέτρα για να ασκηθούν πιέσει ε, στο Ισραήλ, γιατί θεωρούμε ότι για να σταματήσει η βία πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία ειρήνευσης που ξεκίνησε με βάση τη συμφωνία του Όσλο. Θεωρούμε ότι σήμερα δυστυχώς αυτή η διαδικασία είναι ε, ε, παγωμένη, δεν υπάρχει ε, οποιαδήποτε προοπτική να προχωρήσει αυτή η διαδικασία όσο δεν υπάρχει η κατάληξη, της, ο τερματισμός μάλλον της κατοχής και η αναγνώριση ότι, του Παλαιστινιακού κράτους για να λειτουργήσουν δύο κράτη ειρηνικά δίπλα-δίπλα τότε θα συνεχίζονται αυτές οι, οι, οι σκηνές βίας και η μαζική παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως είδαμε να εκφράζεται ε, στη Γάζα. Ε, άρα εκείνο που πιστεύουμε είναι ότι εμείς ε, ως Ευρωκοινοβούλιο πρέπει να στηρίξουμε τη διαδικασία ενηρεύσης αλλά είναι καιρός να μελετήσουμε και μέτρα τα οποία θα πρέπει να στραφούν απέναντι στην κυβέρνηση του Ισραήλ ώστε πρώτα-πρώτα να σταματήσει ο επικισμός που είναι η βασική αιτία ε, που σταμάτησε η διαδικασία ε, να σταματήσουν οι παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στη Γάζα αλλά και στα Παλαιστινιακά εδάφη και την ίδια ώρα βεβαίως να καταδικάσουμε τις όποιες τρομοκρατικές ενέργειες γίνονται από οργανώσεις ή μεμονωμένα πρόσωπα ε, και ε, θεωρώ ότι η έκθεση της κυρία Ντέβης και την ευχαριστούμε γι' αυτό είναι ένα σημαντικό εργαλείο που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ως ε, ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να σταματήσει η βία, να σταματήσει η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να αναγνωριστούν ε, τα δικαιώματα του Παλαιστινιακού λαού, ιδιαίτερα η, η ανακήρυξη και η λειτουργία ενός ανεξάρτητου κράτους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Τώρα θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους. Ο κύριος Πρέδα. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ επίσης την κυρία Ντέιβις για αυτή την παρουσίαση της έκθεσης στα μέλη της Επιτροπής. Βεβαίως, όπως ε, το τόνισε ήδη, λυπούμεθα για το γεγονός του ότι η έκθεση αυτή γίνεται χωρίς καμιά επαφή επιτόπου. Είναι μια έκθεση που δεν έγινε με βάση μια εμπειρία εκεί επιτόπου. Ε, και εξού και κάποια δυναμία ε, της έκθεσης. Εγώ προσωπικά δεν είμαι ε, στρατιωτικός εμπειρογνώμων και νομίζω ότι αυτή του είδους η έκθεση θα πρέπει να εκπονείται κυρίως από την άποψη των ε, στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων οι οποίοι μπορούν να κρίνουν ε, από την άποψη αυτή τι γίνεται. Χωρίς να είμαι εμπειρογνώμων, είδα βεβαίως ένα βίντεο που με εντυπωσίασαν πάρα πολύ, δηλαδή βίντεο που δείχνουν ότι ε, πολίτες της Γάζας βάζανε ε, πολίτες πάνω στις στέγες των σπιτιών που ήξεραν ότι θα μπορούσαν να γίνουν ε, θύματα, θα μπορούσαν να γίνουν στόχοι. Και καταλαβαίνω πολύ καλά τη συγκίνηση της κυρίας Ντέιβι σχετικά με το θέμα αυτό. Είδα αυτή την τρομερή ιστορία με τις σύραγγες που ξεκινούν από την Γάζα και φτάνουν στο Ισραήλ. Και πάλι και εγώ αυτό θα ενδιαφερόμουν για την ε, άποψη των στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων σε σχέση με την έκθεση αυτή. Διότι εμείς που δεν είμαστε στρατιωτικοί δεν μπορούμε βλέποντας εικόνες να εκφέρουμε κρίσεις. Ε, θα ήθελα δηλαδή την ε, εμπειρογνωμοσύνη εμπειρογνωμόνων στρατιωτικών. Ποια είναι η γνώμη τους αυτών που συμβουλευτήκατε. Από πολιτικής απόψεως θα ήθελα να προσθέσω κάτι. Είμαστε το 2015 ε, και γιορτάζουμε τα 40 χρόνια σχέσεις με το Ισραήλ. Και στιγματίζεται συστηματικά. Έχουμε εδώ αυτή την πρακτική στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στιγματίζουμε το Ισραήλ, ξεχνώντας ότι είναι η μοναδική δημοκρατία στη Μέση Ανατολή. Χτες ήδη υπήρξε πρόσθετη ένταση με το θέμα της σήμανσης των προϊόντων, που είναι κάτι το ανόητο από απόψεως εμπορικής και πολιτικής, είναι κάτι το ανόητο είναι μια, αυτή η εξαίρεση που γίνεται και οι Ισραηλινοί αντέδρασαν για αυτήν την κατάσταση η οποία αναφέρεται στα εδάφη και στην πράσινη γραμμή και που δεν, έχει, δεν συμπληρώνεται με τίποτα. Δικαίως οι Ισραηλινοί μας κατακρίνουν για μέτρα χωρίς προηγούμενο. Δεν υπάρχουν τέτοια μέτρα αλλού και δεν έχουμε απάντηση να δώσουμε σχετικά με το θέμα αυτό. Εγώ νομίζω ότι το πραγματικό πρόβλημα όταν πρόκειται για τη Γάζα είναι να έχουμε μια στάση πολιτική για την τρομοκρατική οργάνωση που επικρατεί στη Γάζα. Και αυτό είναι κάπως γελίο να ε, κατακρίνουμε περισσότερο μια δημοκρατία που έχει περισσότερους δεσμούς και κοινά πράγματα με εμάς στην Ευρώπη Δηλαδή μας ανησυχεί περισσότερο το Ισραήλ παρά η Χαμάς. Αυτό είναι το πρόβλημα εδώ και νομίζω ότι έχουμε μεγάλο πρόβλημα πολιτικό από την άποψη αυτή. Ναι, φαίνεται ότι έχουμε πολιτικό πρόβλημα. Κύριο Σπαντσέρη. Όχι, έχουμε ένα πολιτικό πρόβλημα. Είναι προφανές. Εγώ ναι, τονίζω ακόμα περισσότερο τα όσα είπατε. Ναι, υπάρχει πολιτικό πρόβλημα κυρίως ε, από τις διαφορετικές σκοπιές μεταξύ μου και του κυρίου Πρέντα, γιατί υπάρχει το πρόβλημα αντιμετωπίζοντας το από το τέλος και όχι από την αρχή. Το Ισραήλ έχει τεράστια ευθύνη σε σχέση με την ρευτική διαδικασία στα κατεχόμενα και έτσι λοιπόν το τελματώνει η κατάσταση προέρχεται από την εχθρική στάση του Ισραήλ απέναντι στην ερετευτική διαδικασία. Φυσικά, κατόπιν ε, υπάρχουν τεράστιες ευθύνες. Εγώ ευχαριστώ την ε, δικαστή Davis ε, και μπορώ να πω με ειλικρίνη ότι υπάρχει ένα είδος ηρωνίας ε, με την επιχείρηση του Ισραήλ και τον τίτλο το οποίο έφερε. Ουσιαστικά αναφερόταν στην προστασία. Είχαμε 6.000 ενέργειες επιθέσεις και 50 χερσαίες επιθέσεις και είχαμε 1.500 θύματα, το 1 τρίτο ήταν παιδιά. Και όλα αυτά μας δείχνουν ότι έχουν διαπραχθεί από τους Ελληνούς εγκλήματα πολέμου όταν βομβάρδισαν τις κατοικημένες περιοχές ε, στη Γάζα. Και επίσης, ε, βάσει και μιας ε, νομοθεσίας, η οποία θεσπίζει ότι αν συλληφθεί ένας στρατιώτης μπορούν με μέσα άνισα να απαντήσουν οι Ισραηλινοί. Θεωρώ λοιπόν ότι υπήρχαν τεράστιες παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και διαπράχθησαν και κλίματα πολέμου, γιατί οποιαδήποτε επιχείρηση γίνεται θα ε, πρέπει να διαχωρίζει τους στρατιωτικούς από τους μη στρατιωτικούς στόχους. Αυτό δεν έγινε σε καμία περίπτωση. Πρόκειται λοιπόν για μια πολύ σοβαρή κατάσταση. Έτσι λοιπόν τώρα θέλω να ρωτήσω. Έχω παντούτε την ανησυχία όταν μιλάμε για το Ισραήλ ότι κατόπιν φτάνουμε σε ένα συγκεκριμένο σημείο ε, και κατόπιν καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια. Έγινε η έρευνα, είναι αρκετά ξεκάθαρη. Πώς είναι δυνατόν να κλείσουμε αυτό τον κύκλο της ατιμορρησίας. Πώς είναι δυνατόν. Θα έλεγε κάποιος ότι θα έπρεπε να ε, θα πάρουμε μία σειρά μέτρων, όπως παραδείγματο χάρη ένα εμπάργκο όπλων και προς το Ισραήλ και προς τις ένοπλες Παλαιστινικές ομάδες. Όμως θεωρώ ότι θα έπρεπε να σκεφτούμε πάρα πολύ προσεκτικά όλα αυτά τα πράγματα. Αν είναι βέβαια αυτά τα γεγονότα, θα πρέπει η διεθνής κοινότητα να πάρει πάρα πολύ σοβαρά μέτρα, ανεξάρτητα από το πώς μπορεί να αξιολογούμε την Ισραηλινό-Παλαιστινιακή σύραξη. Θα πρέπει να πάρουμε σοβαρά μέτρα γιατί οι δυνάμει επιτόπου και από ό,τι λέω κανένα δεν υπερασπίζεται περισσότερο ένα μέρο από τι άλλο. Αλλά οι δυνάμεις αυτές ε, έχουν αντικειμενικές αποκλίσεις και αν δεν ξεκινήσουμε από αυτή την προϋπόθεση τότε ε, κινδυνεύουμε να μην δούμε ξεκάθαρα τα προβλήματα. Έτσι λοιπόν, μετά από αυτή την εξαιρετική δουλειά που κάνατε με την ε, Εξεταστική Επιτροπή, θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς είναι δυνατόν αυτός ο κύκλος της ατιμορρησίας μπορεί να κλείσει. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ που οργανώσατε αυτόν τον ε, διάλογο και ευχαριστώ την κυρία Ντέιβις που μας έδωσε μια τόσο σημαντική παρουσίαση πολύ δύσκολη. Ξέρω ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να συνοψίσει όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσίαση και για ότι ήσασταν προετοιμασμένοι να συμμετάσχετε σε αυτή τη συζήτηση. Ένα από τα προβλήματα που υπάρχει είναι ότι ε, πολλά πράγματα αναφέρονται, αλλά μετά την έκδοση όλων αυτών των στοιχείων, τη δημοσίευση, τι γίνεται μετά. Δεν ξέρω, εδώ ελπίζουμε στο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι καλώντας σας ε, εδώ θα μπορούσατε ε, να συμβάλλετε εμείς και εσείς ούτως, για το, ούτως ώστε να χρησιμοποιηθεί αυτή η εργασία και να δοθεί συνέσια. Η πρώτη μου ερώτηση είναι, είσαστε δικαστής με ε, μεγάλη εμπειρία και καριέρα σεβαστή. Όταν σας ζητήθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη να κάνετε αυτή την έκθεση, θα είχατε ορισμένες αμφιβολίες αν θα μπορούσατε να το πράξετε ε, και να δώσετε συνέσχεια σε αυτό το σημαντικό θέμα. Είδατε τι συνέβη με άλλες εκθέσεις. Κατά την, η, προηγούμενη έκθεση Gold Report ήταν αξιόπιστη και ε, επέσυρε την προσοχή ε, των πολιτικών. Διαρωτώ ότι και εσείς όταν δεχθήκατε αυτόν τον διορισμό σκεφτήκατε αν θα δοθεί συνέχεια σε αυτήν την έκθεση αν θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά τα πράγματα από ότι με την προηγούμενη έκθεση και ποια είναι η κατάσταση σήμερα βεβαίως εσείς ε, υποβάλατε την έκθεσή σας. Εσείς ε, τι νομίζετε, ποια είναι η τωρινή, σημερινή κατάσταση. Ίσως να μην θέλετε να απαντήσετε ε, σε αυτήν την ερώτηση, αλλά εμεί εκπροσωπούμε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολλές από αυτές είναι μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Ποιο είναι το μήνυμα που εσείς θέλετε να μας διαβιβάσετε σχετικά με την κατάσταση και με την τύχη αυτής της έκθεσης. Μιλήσατε για το τι κάνατε σε σχέση ε, με την αρχή ε, και πολιτικά αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε σε αυτό το κοινοβούλιο και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ε, να μπορούμε να επαναφέρουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τα δύο μέρη Έχουμε βεβαίω ψηφίσματα, αλλά αυτό δεν ξέρω μπορεί να επιτευχθεί. Πρέπει να επιτευχθεί με τον ε, κανόνα, ε, της, ε, του κανόνα δικαίου, του κράτους δικαίου, εάν εμείς οι ίδιοι αγνοούμε αποδείξεις του τύπου που εσείς υποβάλλατε, ε, πώς μπορούμε εμείς ε, να δικαιολογήσουμε τα διάφορα μέρη. Δεν ξέρω αν είναι σχόλιο ή ερώτηση που σας απευθύνω, αλλά δεν ξέρω αν θέλετε να απαντήσετε και πάλι σας ευχαριστώ θερμά για την εργασία την οποία εκπληρώσατε. Λοιπόν, πέρα από πολιτικό πρόβλημα έχουμε και θέμα χρόνου. Μου έχουν ζητήσει οκτώ άτομα το λόγο και επίση θα ήθελα και πρόσωποι από τι πρεσβείε να μπορούν να πάρουν το λόγο, να μπορέσουν να πάρουν το λόγο και να μπορέσει να απαντήσει και η κυρία Ντέιβι. Έτσι λοιπόν, σα παρακαλώ, και ξέρω ότι είναι δύσκολο, να είστε σύντομοι. Παρακαλώ, επόμενο ομιλητή. Eh, ehm. Ευχαριστώ, θα μιλήσω Ολλανδικά. Κυρία Ντέιβις, και εγώ να σας ευχαριστήσω που ήρθατε και μας κάνετε αυτή την παρουσίαση. Σας ευχαριστώ πολύ και για την εξαιρετική εργασία που διεκπαιρεώσατε με τους συνεργάτες σας έτσι ώστε να εξετάσουμε αυτά που συνέβησαν το καλοκαίρι του 2014. Εγώ διάβασα την έκθεσή σας και πραγματικά Πρέπει να σας πω ότι η βία αυτής της σύγκρουσης με σόκαρε. Η λέξη σύγκρουση εξάλλου είναι ορθή. Γιατί εδώ μιλάμε για καταστροφή, για θάνατο. Η Χαμάς και ο Ισραηλινός στρατός τελικά είναι κάποια από τα στοιχεία, μία από τις φάσεις, μία συγκρουση που κρατάει εδώ και πολλά χρόνια μεταξύ των Παλαιστινίων και του Ισραήλ. Μία σύγκρουση η οποία σαφώς και δεν βελτίωσε τίποτα στην περιοχή. Είμαστε υπέρ μιας ειρήνης, δίκαιης και βιώσιμης μεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστίνης και εσείς μιλήσατε για μια δίκαιη λύση αυτό βεβαίως ε, λένε και οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που ζουν στην περιοχή. Εμείς είμαστε υπέρ της προστασίας των δικαιωμάτων και των δύο αυτών εθνών, γι' αυτό και είμαστε κατά της κάθε ε, έκφρασης βίας προς τον άμαχο πληθυσμό και από μέρους των Ισραηλινών αλλά και από μέρους των Παλαιστινίων. Και θεωρούμε ότι βεβαίως το Ισραήλ πρέπει να προσπιστεί τα δικαιώματα των πολιτών τους, αλλά χρησιμοποιώντας ε, ανάλογες, ε, αν θέλετε, ανάλογα μέσα σε σχέση με την απειλή. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ των στρατιωτικών στόχων και του άμαχου πληθυσμού και σε καμία περίπτωση οι πολίτες δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να συνεχίζεται αυτή η σύγκρουση ή για να δικαιολογείται μια τέτοια επέκταση και συνέχιση της βίας. Καταδικάζουμε την ε, πολιτική του Ισραήλ κατά της Λωρίδας της Γάζας, τον αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας και τελικά βλέπουμε ότι αυτοί που πλήττονται, αυτοί που υποφέρουν, αυτοί που βρίσκονται σε μια αδιέξοδη κατάσταση είναι οι άνθρωποι που ζουν στη Λωρίδα της Γάζας. 8 εκατομμύρια Παλαιστίνοι υποφέρουν σήμερα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να βρεθεί λύση και η ερώτηση του κυρίου Χάουιτ είναι πολύ ε, ενδιαφέρουσα για μένα. Πώς πιστεύετε ότι θα δοθεί συνέχεια σε αυτήν την ε, έρευνά σας από τη διεθνή κοινότητα. Γιατί βεβαίως το Ισραήλ προσπαθεί αυτή τη στιγμή να ανταποκριθεί με λογικά επιχειρήματα στις ε, διαπιστώσεις της Εξεταστικής Επιτροπής. Τι ε, προτίθεστε να κάνετε από εδώ και πέρα, γιατί βεβαίως αυτά τα περίφημα rules of engagement είναι εξαιρετικά χαλαρά και σε καμία περίπτωση δεν έχουν επιτρέψει βελτίωση της κατάστασης. Ο κύριος Νόισερ από την Αντιπροσωπή για τη σχέση με την Παλαιστίνη. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Ντέιβις για την έκθεσή της Βεβαίως υπάρχει μια μεγάλη αδυναμία σε αυτήν την ε, έκθεση. Βλέπω δηλαδή το θέμα της επικαιρότητα. Και ακούστηκε ότι εδώ στοχεύουμε το Ισραήλ. Μα το Ισραήλ μονίμως αρνείται να δώσει την οποιαδήποτε πρόσβαση, ακόμα και σε μέλη των αντιπροσωπιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην περιοχή της Γάζας. Αρνείται. Και το είδαμε αυτό πολύ πρόσφατα. Είδαμε πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση επιτόπου όσον αφορά τις άδειε και την πρόσβαση. Και βλέπουμε σε τι αδιέξοδο ζουν αυτοί οι άνθρωποι, χωρίς καμία προοπτική. Δεν χρειάζεται λοιπόν εδώ να συζητήσουμε αν χρειάζεται στρατιωτική εμπειρογνωμοσύνη ή έρευνα. Για κάθε άνθρωπο που προσπασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα ξέρει ότι τόσοι νεκροί, τόσα παιδιά από τον άμαχο πληθυσμό, τόσα θύματα σαφώς και αποτελούν παραβίαση, τουλάχιστον παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και βεβαίως ε, Έχουμε πολλά προγράμματα και σχέδια στη Λωρίδα της Γάζας που στηρίζονται και χρηματοδοτούνται από τον Ευρωπαίο φορολογούμενο. Και είναι πολύ σημαντικό ε, όλη αυτή η ανθρωπιστική βοήθεια, όλη αυτή η προσπάθεια να προχωρήσουν και να συνεχιστούν αυτά τα προγράμματα που έχουν πληγεί από αυτά που συμβαίνουν εκεί, να συνεχιστούν. Είναι προγράμματα για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, νερού και βλέπουμε ότι έχουν καταστραφεί αυτές οι υποδομές από τις ε, Ισραηλινές αρχές. Οι εκτιμήσεις σας λοιπόν είναι πολύ σημαντικές για μας. Εμείς σαν Ευρωπαϊκή Ένωση τι μπορούμε να κάνουμε και για να σταματήσει αυτή η στόχευση προς το Ισραήλ κάνουμε μια έκκληση προς αυτούς να συνεργαστούν. Το θέμα, παραδείγματο χάρη των ε, ετικετών και της σήμανσης των προϊόντων που προέρχονται από τα καταχώμενα είναι κάτι το οποίο δεν είναι αυτοσκοπός. Πρέπει όμως να υπάρξει μία αλλαγή στάσης, γιατί βλέπουμε ότι οι ακραίες δυνάμεις του Ισραήλ συνεχίζουν να καθορίζουν την πολιτική. Ο κύριος Αντάκτουσον. Eh, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Ντέιβις για την παρουσίασή της. Όλοι, όλοι έχουμε πραγματικά σοκαριστεί όταν βλέπουμε τις σημαντικές επιπτώσεις αυτής της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης. Εγώ έχω πάει στην Λωρίδα της ε, Γάζας, έχω πάει και στο νότιο Ισραήλ, όπου είναι εμφανής ε, ο αντίκτυπος αυτής της μακροχρόνιας σύγκρουσης. Στην έκθεσή σας υπάρχει παρόλα αυτά κάτι, μια πολύ λεπτομερής ανάλυση των αιτιών ε, αυτής της συνεχιζόμενης σύγκρουσης και αυτό που θα ήθελα εδώ να σας πω είναι ότι γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία καθοδηγείται από μια τρομοκρατική οργάνωση, την Χαμάς, που όπως ξέρετε θεωρεί ότι το Ισραήλ θα πρέπει να εξαλειφθεί από προσώπου γης. Βεβαίως βλέπουμε ότι η Χαμάς με την διεύθυνση την Παλαιστινιακή κάθε χρόνο συνεχίζει μια προπαγάνδα κατά του Ισραήλ, μια αντισημιτική πολιτική με μια σειρά όρους και προϋποθέσεις που δεν μπορεί παρά να επιδεινώσουν την κατάσταση επιτόπου. Εάν κανείς δεν αλλάξει αυτήν την προσέγγιση, δεν υπάρχει περίπτωση να κατανοήσουμε αυτά που συμβαίνουν στη λωρίδα της Γάζας. Τώρα, όσον αφορά το καλοκαίρι του 2014, αυτό που συνέβη εκεί σαφώς και οφείλεται και στις διαρκείς απειλές κατά του Ισραήλ. Είναι δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο είναι υποχρεωμένο το Ισραήλ να προστατεύσει τους πολίτες του, να προστατεύσει τον λαό του από όλες τις εξωτερικές απειλές. Και βεβαίως βλέπουμε ότι το Ισραήλ αυτή τη στιγμή επίσης βρίσκεται σε μια αδιέξοδη κατάσταση. Πρέπει να αντιμετωπίσει τις απειλές της διεθνούς τρομοκρατίας, αυτήν την προπαγάνδα, την αντισημιτική και μία σειρά δραστηριοτήτων που μειώνουν τις προοπτικές ε, για μία μελλοντική ειρηνική συνύπαρξη στην περιοχή. Επαναλαμβάνω ότι το διεθνές δίκαιο δίνει δικαίωμα στο Ισραήλ να αμυνθεί, να προστατεύσει τον πληθυσμό του. Και μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κατανοήσουμε αυτά που συμβαίνουν εκεί, ιδιαίτερα αυτά που συνέβησαν το καλοκαίρι του 2014. Όλοι ξέρουμε ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η βία, να σταματήσει η αιματοχυσία στην περιοχή, να υπάρξει μια λύση με ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος και ένα Ισραήλ χωρίς συνεχιζόμενες απειλές και αντισημιτική προπαγάνδα. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω την άποψή σας γιατί στην έκθεση αυτή συνεχίζουν να παρουσιάζονται στοιχεία τα οποία κατά τα άλλα δεν συζητούνται και δεν βρίσκονται στην διεθνή συζήτηση. Συγγνώμη που επιμένω, αλλά είναι θέμα σεβασμού και στους υπόλοιπους συναδέλφους. Έχουν ζητήσει πολύ το λόγο και θεωρητικά στις 11 θα έπρεπε να τελειώσουμε. Αν θέλετε να απαντήσει και η κυρία Ντέβης, θα πρέπει να είστε πιο σύντομοι, διαφορετικά θα μπορέσει να απαντήσει ο κύριος Οστρεβίτσιος. Ευχαριστώ, δεν άκουσα καλά το όνομά μου. Κυρία Ντέιβις, θέλω να σας ευχαριστήσω για την έκθεσή σας. Αυτή ε, δεν ήταν ε, μια απλή έκθεση. Από ό,τι κατάλαβα ήσασταν πολύ συγκινημένοι όταν ε, μας κάνατε όλη την περιγραφή της διαδικασίας. Βέβαια, από ό,τι κατάλαβα δεν μπορέσατε να μεταβείτε εκεί και να τα δείτε με τα ίδια σας τα μάτια. Έχω βέβαια κάποια σχόλια το Ισραήλ, όπως ε, και κάθε κράτος έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα και να διασφαλίσει την ασφαλεία των πολιτών του. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό, να γνωρίσουμε το δικαίωμα αυτό και για τον εαυτό μας. Αν ε, η Χαμάς ε, συνεχίζει να αναφέρει ότι είναι αποφασισμένη να εξελίψει το Ισραήλ, δεν θα υπάρχει ασφάλεια, το γνωρίζουμε αυτό. Έχετε δίκιο ότι μεταξύ των Παλαιστινίων θεμάτων οι περισσότεροι ήταν άμαχοι. Ναι, είναι λογικό αυτό, γιατί και η Χαμάς χρησιμοποιεί ε, ανθρώπους ως ασπίδες Νομίζω ότι αυτό το κάνει εκ προθέσεως και δεν είναι ανθρώπινο. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να αποφύγουμε την ύπαρξη θυμάτων σε όλες τις πλευρές, όλα αυτά. Υπάρχει ένας πόλεμος, ε, ο οποίος ε, συνεχίζεται και είναι δηλωμένος και αδήλωτος πόλεμος. Έχουμε και τα μαχαιρώματα, άνθρωποι μαχαιρώθηκαν στο δρόμο, άμαχοι, Όλα αυτά είναι εικόνες ε, του 21ου αιώνα. Πρόκειται για εκδηλώσεις νέων τρομοκρατικών φαινομένων. Και έχω μια ερώτηση. Στις τελευταίες παραγράφους της εκθεσής σας ε, είπατε ότι υπάρχει απάντηση, ότι ελπίζετε ότι θα υπάρχει απάντηση και από το Ισραήλ και από την Παλαιστίνη υπήρξε τέτοια απάντηση. Μπορείτε να μας πείτε ποια ήταν αυτή, η κυρία Πόστ. Eh, Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την παρουσίαση της έκθεσης. Εγώ είχα μια ερώτηση να θέσω, αλλά αφού άκουσα τα όσα λέχθηκαν από τους συναδέλφους, θα ήθελα να σχολιάσω κάτι άλλο. Θα ήθελα να αρχίσω απαντώντας τα όσα είπα, ελέγχθηκαν. Είναι μια έκθεση που προέρχεται από την προοπτική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεν είναι κάτι που θα πρέπει να το συνδέσουμε με τους στρατιωτικούς. Πρόκειται για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό είναι το θέμα μας ε, για τα παγκόσμια ανθρώπινα δικαιώματα ε, με βάση από έχουν θεσπιστεί από το 1948 μετά τον πόλεμο ε, και τότε δημιουργήθηκε και το κράτος του Ισραήλ. Η έκθεση δεν θα έπρεπε να δικαιολογεί την βία που υπάρχει σε κατάσταση διένεξης ανεξάρτητα με τα όσα μιλάμε εδώ. Μιλάμε για το Δαβίδ και το Γολιάθ εδώ. Δεν θα έπρεπε ε, να λέμε ότι αυτό συμβαίνει, αυτό συμβαίνει εκείνο, αλλά να εστιαστούμε ε, πάνω σε συγκεκριμένα πράγματα που περιγράφονται, πώς υπάρχουν παραβιάσεις ε, σε θέματα κοινών διακηρύξεων, πώς δεν υπάρχει ευθύνη σε επίπεδο διεθνούς κοινότητας και θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα της ευθύνης, της λογοδοσίας του Ισραήλ και της διεθνούς κοινότητας και το τι συμβαίνει στις σχέσεις με τη Χαμάσα. Ένα άλλο θέμα που τίθεται, το άρθρο 30, ε, ήταν αρκετά σαφές τι μπορούμε να κάνουμε ούτως ώστε συγκεκριμένα να μπορούμε να έχουμε μια πραγματική εφαρμογή, μια πραγματική αποτελεσματικότητα. Τι μέσα διαθέτουμε. Θα πρέπει και πάλι να συναντηθούμε, να συμφωνήσουμε για να δούμε πόσα θα πρέπει αυτή η διακήρυξη, η δήλωση ε, να υλοποιηθεί, πώς ε, να ενισχύσουμε τα δικαιώματα των ανθρώπων, των ατόμων. Τι συμβαίνει στην Ευρώπη και τι συμβαίνει εκτός Ευρώπης. Βλέπω ότι η διεθνής κοινότητα αρνείται τη συνεργασία συστηματικά για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις παγκόσμιες προκλήσεις. Ένα άλλο θέμα που τίθεται είναι μπορούμε ε, να θεωρήσουμε ως αρχή ότι η Γάζα είναι ασφαλές έδαφος. Ο κύριος Γκαρίκια και ο κύριος Τέιλορ έχουν ζητήσει το λόγο. Με αυτή τη σειρά παρακαλώ. Θα ήθελα να πω ότι η κατάσταση στην ε, Γάζα αλλά και στο Ισραήλ είναι αποτέλεσμα πολέμου. Βλέπετε πόσα παιδιά έχουν μείνει ορφανά και ε, το θέμα αυτό είναι αυτονόητο, δεν, δεν πρέπει να συζητήσουμε γι' αυτό. Το θέμα είναι όμως ότι κάποια παιδιά χρησιμοποιούνται σαν ασπίδες και θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο και δεν ξέρω πώς μπορεί κάποιος από το Ισραήλ να ξεκαθαρίσει και να διακρίνει αν κάποιος πρόκειται κάποιος νέος που είναι απέναντί τους είναι στρατιώτης, ασπίδα ή ένα απλό παιδί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η Χαμάς βεβαίως έχει εκλεγεί δημοκρατικά και απειλεί, απειλεί την χώρα του Ισραήλ, το κράτος του Ισραήλ με πλήρη εξάλληψη. Για μας αν θέλετε τους Γερμανούς αυτό είναι κάτι το απαράδεκτο. Είναι πολύ δύσκολο να το δεχτούμε. Όταν μιλάμε τώρα για το δικαίωμα, αν θέλετε, της εγκατάστασης. Ξέρετε πολύ καλά ότι εδώ δεν πρόκειται για κάτι το οποίο μπορεί να συμβαίνει και αλλού στον κόσμο, στην Αφρική ή κάπου αλλού. Εδώ ουσιαστικά αν θέλετε πρόκειται για μια ε, κατάκτηση η οποία δεν μπορεί να θεωρηθεί ε, λάφυρο πολέμου. Μιλάμε για κάτι πολύ συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη πολιτική. Και όλα αυτά τα σπίτια, όλες αυτές οι οικοδομήσεις, οι κατοικίες ε, και όλη αυτή η πολιτική επικισμού έχει μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική. Δεν έγινε από τη μία μέρα στην άλλη. Πρόκειται λοιπόν για πόλεμο. Πρόκειται για ένα πόλεμο που πραγματικά απειλεί το Ισραήλ μονομερός με πλήρη εξάλληψη. Και κοιτάξτε το μέγεθος του Ισραήλ. Κοιτάξτε πόσο μικρό είναι το Ισραήλ. Πόσο μικρό είναι. Και είναι πολύ σημαντικό να είμαστε προσεκτικοί και να κατανοήσουμε τις πραγματικές διαστάσεις αυτού του προβλήματος. Εμείς θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε εδώ γιατί αφήσαμε να υπάρξουν στο Ιράκ 100.000 νεκροί. Θα πρέπει να εξηγήσουμε γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας εξοπλισμών, γιατί εκατοντάδες παιδιά τα οποία ζουν σήμερα σε προσφυγικούς καταβλισμούς ε, γύρω από τη Συρία. Όλα αυτά θα πρέπει να τα συνειδητοποιήσουμε για να δούμε πού είναι και η δική μας ευθύνη και ενοχή. Τέιλορ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω την κυρία Ντέιβις. Ήταν πολύ δύσκολο να διεκπαιρεωθεί αυτή η εργασία και να την παρουσιάσει εδώ. Έχω δύο ερωτήσεις. Θα πρέπει όμως να σχολιάσω κάποια από αυτά που ακούστηκαν εδώ όσον αφορά αυτή τη σύγκρουση μεταξύ Παλαιστίνης και Ισραήλ. Βεβαίω, το Ισραήλ έχει δικαίωμα να αμυνθεί. Έχει δικαίωμα αυτό Όμως ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά το Ισραήλ. Θα πρέπει σαφώς να ακολουθείτε και από κάποιες αναλήψεις ευθυνών. Ε, βλέπουμε σήμερα με τον αποκλεισμό της Γάζας, με την πολιτική τοπικισμού, με τις διάφορες συλλήψεις και κρατήσεις, και κυρίως τις, ε, τα πλήγματα κατά του ομάχου πληθυσμού. Όλα αυτά που συμβαίνουν, αν θέλετε, στη Γάζα είναι ε, μια τιμωρητική προσέγγιση και πολιτική κατά των πολιτών αυτής της περιοχής. Αναρωτιέμαι λοιπόν, σας στήριξε καθόλου η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτόπου εκεί στην Παλαιστίνη, οι αντιπροσωπείες. Νιώθετε ότι τα κράτη-μέλη κάνουν αυτά που θα έπρεπε να κάνουν για να σας στηρίξουν. Τι μπορούμε να κάνουμε για να σας στηρίξουμε καλύτερα και να σας βοηθήσουμε στην αποστολή που έχετε αναλάβει. Και η δεύτερη ερώτηση, νομίζω δεν είμαι ο μόνος που την κάνει εδώ, μία από τις συστάσεις σας, στην οποία εντοπίζετε την έλλειψη υλοποίησης συστάσεων που έχουν βεβαίως ε, υποβληθεί από προηγούμενες διερευνητικές εξεταστικές επιτροπές των Ηνωμένων Εθνών. Τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα για να υλοποιηθούν πραγματικά αυτές οι συστάσεις. Ευχαριστώ. Συγγνώμη που σας βιάζω τόσο, αλλά θα ήθελα να δώσω το λόγο στην ε, κυρία Ντέιβις για να προσπαθήσει να απαντήσει στις ε, πολυάριθμες ερωτήσεις που κάνατε και να δώσουμε και το λόγο στους εκπροσώπους από την Πρεσβή της Βελίλα και την Παλαιστίνη. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Έχω μια μακρά σειρά ερωτήσεων που βασικά είναι περισσότερες ρητορικέ διότι δεν μπορώ εγώ να τις απαντήσω διότι δεν είμαι πολιτική εκπρόσωπος. Απλώς κάνω τη δουλειά μου όσο την έκανα όσο καλύτερα μπορούσα επικεφαλής της Επιτροπής αυτής και εκπώνησα ε, την έκθεση. Ε, βεβαίως ο Γάλλος εκπρόσωπος εδώ ε, ε, ρώτησε αν θα έπρεπε ε, να εμπλακούν και στρατιωτικοί εδώ στην έκθεση. Δεν μπορώ να πω ότι διαφθονώ. Ίσως θα ήταν καλύτερα αν είχαμε ε, κάποιον στην Επιτροπή. Αυτή την ερώτηση πρέπει να τη θέσετε σε αυτόν που ε, διόρισε την και συνέθεσε την Επιτροπή. Αυτή ίσως θα ήταν χρήσιμο να είχαμε κάποιον στην Επιτροπή που να ήταν στρατιωτικός εμπειρογνώμων. Βεβαίως είχαμε και έναν εμπειρογνώμονα στρατιωτικό που είχε ε, πρακτική εμπειρία επιχειρησιακή μιας δυτικής δύναμης και το άτομο αυτό μπόρεσε να μας δώσει συμβουλές εμπειρογνώμονα σε σχέση με την εξέταση του θέματος. Αυτό μόνο μπορέσαμε να κάνουμε. Γι' αυτό είχαμε λοιπόν αυτήν την εμπειρογνωμοσύνη για τα μέλη της Επιτροπής. Επίσης πήραμε συνέντευξη από πολλούς εμπειρογνώμονες στρατιωτικούς, πολλούς από το Ισραήλ και προσπαθήσαμε κατά κάποιο τρόπο να καλύψουμε την έλλειψη εμπειρογνωμοσύνης. Βεβαίως, η στρατιωτική άποψη δεν είναι σχετική, ε, λένε πολλοί, αλλά εγώ νομίζω ότι είναι σχετική εφόσον πρόκειται για πόλεμο, αλλά βεβαίως εστιαστήκαμε κυρίως στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και πάρα πολλές από τις περιπτώσεις που εξετάσαμε και αυτό είναι που καθιστά δύσκολο να πούμε ότι αυτό πράγματι συνέβη, πράγματι έγινε αυτό. Βεβαίως δεν είναι τόσο σαφή τα πράγματα, ε, κυρίως το ανθρωπιστικό δίκαιο, κυρίως αν δεν έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζεστε για να εκφέρετε κρίσεις. Ε, ποια ήταν η επιλογή όπλων, τι πράγματα σκεφτήκατε ε, πρώτου να, ρίξετε αυτή τη βόμβα τόσων τόνων. Βεβαίως δείχνουμε τι ε, κατά τη γνώμη μας είναι ε, πού είναι τα προβλήματα ούτως ώστε αν κάποιος έχει τα μέσα, έχει την πολιτική στήριξη και ότι χρειάζεται να τα, να τα θέσει στη διάθεση ούτως ώστε να γίνει μια πραγματικά επαγγελματική έρευνα. Εμείς δεν τα είχαμε αυτά τα μέσα, δεν είχαμε αυτούς τους πόρους, δεν πρόκειται να μιλήσω ε, για τα διάφορα ε, θέματα αυτά. Αυτό είναι θέμα ε, των Ηνωμένων Εθνών. Είχαμε πολλές δύσκολες περιπτώσεις και κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Ε, δεν πρόκειται να εκτιμήσουμε τον Ταβί και τον Γολιάθ, να δούμε θέματα ηθικής. Είχαμε θέματα αρχές διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όλα αυτά τα θέματα ασχοληθήκαμε σχετικά με τα μέρη που βρίσκονται εκεί και, και κρίναμε με βάση αυτά τα πρότυπα, αυτούς τους κανόνες. Τι θα συμβεί ε, με την έκθεση, θα μπει σε κάποιο ράφι νομίζω, εκτός αν κάτι αλλάξει στην όλη δυναμική σε αυτήν την περιοχή. Ε, όταν είδα ότι ο πρόεδρος Ομπάμα μάλλον εγκατέλειψε την μάχη δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Ελπίζω ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην έχει εγκαταλείψει την προσπάθεια να κάνει, να μην φυστεί καμιά προσπάθεια για να κάνει ό,τι χρειάζεται σχετικά με τα θέματα αυτά. Θα πρέπει να υπάρχει μια διαπραγμάτευση που θα οδηγήσει στην ειρήνη, ασφάλεια για το Ισραήλ, αυτοδιάθεση ε, για τους Παλαιστίνιους, ε, να μάθουν όλοι ο ένας κοντά στον άλλον και ε, να δούμε τι, πώς θα μπορούσε να υπάρξει μια συμφωνία, αν υπάρχει πολιτική βούληση στην ε, περιοχή. Ε, δεν είναι θέμα για, έναν, για μια συνταξιούχο δικαστή. Δεν μπορώ να σας πω εγώ προσωπικά τι θα ήθελα να συμβεί. Αυτό που με απασχολεί και με ανησυχεί είναι η ατιμορρησία και θα πρέπει και νομίζω ότι το Ισραήλ έχει κάνει προόδους βάζοντας πληροφορίες στο διαδίκτυο. Θα πρέπει να παρακολουθούμε με προσοχή. Άκουσα ότι θα μπορούσαν να γίνουν ε, σύλληψεις ε, στην Γάζα από τις αρχές ε, είδα ένα άρθρο πριν μερικές μέρες ε, στη New York Times και πάλι θα πρέπει να παρακολουθούμε και να ασκήσουμε πίεση στις ε, διάφορες ομάδες. Διότι το καλύτερο πράγμα είναι ίσως να κάνουν τις έρευνες οι διάφορες ομάδες. Αλλά πρέπει να εξετάσουμε τα πράγματα και διάφορες ορισμένοι έχουν κληθεί για να βοηθήσουν ε, στην όλη έρευνα του θέματος και αυτή η εμπειρία θα ήταν διαφορετική από την προηγούμενη εμπλοκή μου. Ήμουνα ε, για, ε, ασχολήθηκα με την έκθεση Goldstein, με το τι έγινε με την πρώτη έκθεση, με τις συστάσεις, αν οι συστάσεις αυτές είχαν εφαρμοστεί, είχαν υλοποιηθεί. πήγα στην Γάζα το 2010 Ξέρω πολύ καλά την αθλειότητα που υπάρχει, την πτώχεια που υπάρχει σε αυτήν τη λωρίδα γης. Αλλά βεβαίως δεν μπορέσαμε να πάμε αυτή τη φορά και αυτό είχε να κάνει τόσο με την κατάσταση ασφαλείας στο βόρειο μέρος του Σινά και δυστυχώς δεν μπορέσαμε να πάμε και κάναμε ό,τι μπορούσαμε με τις περιστάσεις που είχαμε. Ε, δεν μπορέσαμε να κάνουμε περισσότερα από αυτά που μπορούσαμε λόγω των περιορισμών που είχαμε. Και αν θα μπει σε ράφη αυτή η έκθεση, τι θα γίνει ε, τελικά. Νομίζω και, και νομίζω ότι όταν διαβάζω μερικές μαρτυρίες μαρτύρων ε, παρουσιάζουν τις φωνές τους. Δεν μπορώ να σας πω τι θα γίνει. Πηγαίνουν εκεί, ε, ε, λένε αυτή τη φορά θα είναι διαφορετικό αν σας μιλήσουν τα άτομα αυτά. Το θέμα είναι ότι καταγράφετε όλα, έχετε τις φωνές τους στην έκθεση και κάποια μέρα όταν κάποιος θα έχει τα μέσα θα μπορέσει ίσως ε, να, ε, να πάρουν τα πράγματα την οδό της δικαιοσύνης, να γίνουν έρευνες, να γίνουν ανακρίσεις, να γίνουν διώξεις. Ελπίζουμε να φτάσει αυτή η στιγμή. Ευχαριστούμε πολύ. Οι εκπρόσωποι των πρεσβειών θα ήθελαν να μιλήσουν. Θέλετε το λόγο. Μόνο τρία λεπτά μπορώ να σα δώσω. Λυπάμαι, αλλά έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Σα παρακαλώ, προσπαθήστε να είστε σύντομοι. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Βελερτάλ, που είναι υπουργό σύμβουλο τη Πρεσβεία του Ισραήλ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να τονίσω ότι εμείς ε, σεβόμαστε τη Μερή Ντέιβις και τη θέση της ως πρόεδρο της Ανεξάρτητης Εξωτικής Επιτροπής για τη σύραξη στη Γάζα για την προθυμία της να ακούσει και τα δύο πλευρά, ε, έχοντα κατά νου και τα διλήμματα που έχει να αντιμετωπίσει το Ισραήλ. Η εντολή δόθηκε στην κυρία Ντέιβις από το ε, Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΙΕ. Πρόκειται για μια διεθνή αρένα που έχει ε, θέσει συγκεκριμένη ατζέντα κατά του Ισραήλ και επικεντρώνεται στην ισραηλο διαμάχη. Τα τελευταία εννέα χρόνια το Συμβούλιο έχει ε, δημοσιεύσει περισσότερα ψηφίσματα κατά του του Ισραήλ από ό,τι για τον υπόλοιπο κόσμο ε, οι μουσουλμανικές χώρες ψηφίζουν κατά του Ισραήλ. Ε, η κυρία Ντέιβις δεν ελέγχει αυτό το συμβούλιο τι θα κάνει με την έκθεση αυτή. Ως προς την έκθεση ε, είναι απαραίτητο να δούμε τις επιχειρήσεις υπό δύο μορφές. Ε, καταρχήν σε σχέση με τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει το Ισραήλ, όχι μόνο στη Λορδία της Γάζας αλλά και στη Δυτική Όχθη. Και δεύτερον, το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο ε, δεν αντιμετωπίζει ένα μικρατικό φορέα όπως η Χαμάς, αλλά ουσιαστικά υπάρχουν κάποια πρότυπα που εφαρμόζονται διεθνώς. Τώρα λοιπόν πώς προσεγγίζουμε ε, κάποιες τρομοκρατικές οργανώσεις ή αποτυχημένα κράτη όπως η Συρία και το Ιράκ. Εμείς ε, ελπίζουμε ότι ε, θα μπορέσει ε, η Επιτροπή να ασχοληθεί και με άλλες περιπτώσεις όπως τη Δεν κάνει τίποτα όμως, δεν υπάρχει καμία έρευνα ούτε καν καταδίκες. Το κράτος του Ισραήλ έχει εσωτερικούς νομικούς μηχανισμούς και στρατιωτικούς και μη στρατιωτικούς που ε, ουσιαστικά αντιμετωπίζουν καταγγελίες παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτό αντικατοπτρίζεται στην έκθεση της δικαστού. Στην περίπτωση του Ισραήλ κάνουμε περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα, ακόμη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε καταγγελία ε, που υποδηλώνει ότι υπάρχει παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, εξετάζεται από τους αρμοδίους. Αυτές οι έρευνες βασίζονται σε μαρτυρίες από ε, στρατιώτες του Ισραήλ αλλά και από Παλαιστινίους που ήταν μάρτυρες στα περιστατικά αυτά και ενώ εφαρμόζεται πλήρως το σύστημα, το σύστημα του Ισραήλ πρέπει να ρωτήσουμε ποια ήταν η εμπειρογνωσύνη στην οποία βασίστηκε η έκθεση αυτή. Έχουμε κάποιες αμφιβολίες. Το κράτος του Ισραήλ συνεχίζει να σέβεται τα διεθνή πρότυπα του διεθνούς δικαίου και έχει παρουσιάσει στην κυρία Ντέβις όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Ε, σέβεται το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο μία αντιπροσωπεία ε, δέκα στρατηγών ε, με επικεφαλής τον Κλάου Σνάουμεν που επισκέφθηκε τον Ισραήλ κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ε, έδρασαν στα πλαίσια του δικαίου και ουσιαστικά σεβάστηκαν την αναλογικότητα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πρεσβευτής του, του της Παλαιστίνης, με συγχωρείτε, έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ πολύ, κυρία Δικαστέ, για την έκθεσή σας που μας γίνησε ιδιαίτερα. Ευχαριστώ πολύ και για την πρόεδρο της Επιτροπής εδώ που μας δίνει το λόγο. Σκοπός μας δεν ήταν να παραστούμε. Δεν είχε νόημα να πάρουμε το λόγο και να πούμε κάτι που σαφώς αφορά την Παλαιστίνη. Αλλά όταν ακούω την εκπρόσωπο της ε, πρεσβείας του Ισραήλ που πραγματικά αναφέρεται στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από μέρους του Ισραήλ, παίρνω το λόγο για να πω ότι μακάρι, αυτό είναι κάτι που με χαροποιεί ιδιαίτερα. Ακούω ότι είναι κατά της ε, πολιτικής ε, διακρίσεων που έχει ξεκινήσει από το Ισραήλ και έχει σαν θύματα 1500 παιδιά Παλαιστίνιους άμαχους, κάτι που συνεχίζεται με πολλά θύματα. Επίσης, αναφερθήκατε στην κατοχή από μέρος του Ισραήλ που έχει ξεκινήσει το 1948. Αν οι συνάδελφοι από το Ισραήλ επικρίνουν αυτά τα φαινόμενα, σαφώς θα πρέπει να επικρίνουν και την πολιτική κατασκευής επικιών από μέρους του Ισραήλ, κάτι που συνεχίζεται και βεβαίως Είναι πολύ σημαντικό επίσης να αναφερθούμε και στις ε, αποφάσεις ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίες έχουν υποστηριχθεί από 28 διαφορετικές κυβερνήσεις κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να λέμε ότι είναι ανόητες. Διαβάστε σας παρακαλώ πολύ αυτή την απόφαση, διαβάστε επίσης την θέση της διεθνούς κοινότητας είστε μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα πρέπει να γνωρίζετε το διεθνές δίκαιο, θα πρέπει να ξέρετε ότι έχουν χαρακτηριστεί σαν παράνομες αυτές οι επικίες και ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να τις δεχτούμε. Πρόκειται για παράνομες κατασκευές Σε κάθε περίπτωση αυτά που γίνονται σήμερα δεν αρκούν σε μας στους Παλαιστίνιους. Χαιρόμαστε που η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει φιλική στάση προς την ε, Παλαιστίνη, αλλά δεν ζητάμε φίλους, ζητάμε απλώς να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο. Κάνουμε μια έκκληση όχι προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη, αλλά λέμε ότι πρέπει να είστε πιστοί στην προάσπιση των δικαιωμάτων. Ε, ολοκληρώνω, ολοκληρώνω. Δεν θα επανέλθω στο θέμα συζήτησης της σημερινής ε, παρουσίασης. Αλλά πραγματικά ευχαριστώ πολύ την ε, κυρία Δικαστή και την ευχαριστώ λέγοντας ότι μας αρκεί η έκθεσή της για αυτή την έκθεση. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό που μπορεί να βγάλουμε σαν συμπέρασμα είναι ότι δεν μπορεί ε, να δολοφονούνται παιδιά, να βομβαδίζονται νοσοκομεία, να βομβαδίζονται σχολεία και εμεί να ψάχνουμε να δούμε αν πραγματικά είναι παραβίαση ή όχι ανθρωπίνο δικαιωμάτων. Είναι εξόφθαλμα εγκλήματα. Και μπορούμε βέβαια να τα και σωστά τα χαρακτήρισε η κυρία Ντέβη εγκλήματα πολέμου και εδώ είναι που εμεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Το δεύτερο, επειδή άκουσα τη φράση εδώ σε αυτή την αίθουσα να μιλούμε για αντισημιτισμό. Όταν καταγγέλνουμε εγκλήματα δεν είναι αντισημιτισμό. Τα εγκλήματα και την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων την καταγγέλνουν δεκάδε, εκατοντάδε χιλιάδε Ισραηλινοί. Είναι και αυτοί αντισημίτε. Ε, γιατί στο τέλο τη ημέρα ε, θα ξεχάσουμε ποιο είναι το νόημα. Και, και τελειώνω με το εξή. Αυτό που χρειάζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δράση. Δράση για να τερματιστεί η παραβίαση ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να σταματήσουν να δολοφονούνται παιδιά στους δρόμους, να σταματήσει ο επικισμός και να βοηθήσουμε να συμβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να υπάρξει ειρήνη. Και η ειρήνη δεν μπορεί να υπάρξει στη Μέση Ανατολή όσο υπάρχει κατοχή. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Θέλετε να πείτε κάτι τελευταίο? Απλώς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την προσοχή σας και ελπίζω ότι θα έχετε ακούσει τις φωνές των ανθρώπων και στο Ισραήλ και στα κατεχόμενα εδάφη, τα Παλαιστινιακά που καλούν τους ηγέτες τους αλλά και όλους εσάς να φέρετε μια πραγματική και μακροπρόθεσμη ειρήνη και για τις δύο πλευρές και την ύπαρξη δύο κρατών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λέει πρόεδρος, ξέρετε, είναι μια δύσκολη συζήτηση αυτή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι πολύ σημαντικό να ακούμε μια τόσο έντιμη φωνή. Πραγματικά είναι μεγάλη ικανοποίηση για μας να σας ακούμε. Ολοκληρώνουμε λοιπόν εδώ αυτό το σημείο. Vamos Για να περάσουμε στο επόμενο σημείο. Όσοι θέλετε να εγκαταλείψετε την αίθουσα, παρακαλώ να το πράξετε. Θα περάσουμε στο θέμα της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο ότι ξέρετε ότι η αμφισβητούμενη εκλογή του Πρόεδρου Κουρουζίσα για μια τρίτη θητεία προκάλεσε μια πολιτική και κοινωνική και ανθρωπιστική καταστροφή. Σήμερα είχαμε καλέσει στην Επιτροπή μας τον ε, κύριο Πιέρ Κλαβέρ Μπονίμπα, έναν ε, από τους πιο διάσημους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπουρούντι για να καταθέσει μαρτυρία στην Επιτροπή μας για την κατάσταση στη χώρα του. Ο Πιέρ Κλαβέρ ε, είναι υπό ε, θεραπείας νοσοκομείο στο Βέλγιο γιατί του επιτέθηκαν. Ε, ήταν πολύ σοβαρά, τώρα είναι λίγο καλύτερα. Και περασμένη Παρασκευή ο 25χρονος γιος του δολοφονήθηκε στην Μπουζουμπούρα και πριν είχε δολοφονηθεί και ο γαμπρός του. Το πτώμα του γιού του βρέθηκε κατόπιν σύλληψής του από την αστυνομία και Λόγω του πένθους, ο κύριος Κλεβέρ ε, δεν μπορεί να παρευρεθεί εδώ, λυπούμαστε πάρα πολύ. Την κατάσταση θα μας την περιγράψει συνέχεια συνέχεια συνάδελφος. Είναι καταστροφική η κατάσταση. Η κυβέρνηση του Μπουρούντι μπροστά στην κατάσταση αυτή εξέδωσε ένα τελεσίγραφο στον ίδιο του τον πληθυσμό και αυτό το μόνο που έκανε ήταν να επιδεινώσει την αίσθηση του φόβου και της ανασφάλειας ε, που διατρέχει τη χώρα. Φοβούμαστε ότι η χώρα ολισθαίνει προς εμφύλιο και Γνωστοποίησαμε αυτή την ανησυχία μας και στην είπατε πρόσωπο, αλλά και στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε καλέσει εδώ διάφορους εμπειρογνώμονες που θα μπορούσαν να μας περιγράψουν την κατάσταση, πώς έχει σήμερα αυτή τη στιγμή καταρχήν. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Βερκούλο. Ευχαριστώ. κυρία Πρόεδρε, είμαι Βιρκουλό. είμαι Διευθυντής για την Κεντρική ε, Αφρική στο International Crisis Group. Η International Crisis Group εργάζεται για το Μπουρούντι από την εποχή ε, του 1998, την εποχή του εμφουλίου πολέμου και από τότε δεν έπαψε να παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης στο Μπουρούντι, είτε για την ε, Συμφωνία της Αρούσα, την υλοποίηση και από τις τελευταίες εκλογές. Τώρα μπήκαμε στην τρίτη φάση της κρίσης στο Μπουρούντι. Η πρώτη φάση είχε αρχίσει το 2014 με μια διένεξη εκλογική και την ασυμφωνία για τις διάφορες προετοιμασίες εκλογικές μεταξύ των εμπλεκομένων ενδιαφερομένων μερών. Η δεύτερη φάση άρχισε τον Απρίλιο φέτος με ταραχές στους δρόμους για τον πρόεδρο Μπουρουντιζά και ε, σαφής αντιπαράθεση με αφενός ε, την κοινωνία των πολιτών, την αντιπολίτευση ε, και την νεολαία στη Μπουζουμπούρα και από την άλλη πλευρά την εξουσία και στη δεύτερη αυτή φάση άρχισε η κρατική βία. Από το θέρος άρχισε και από την ε, επανεκλογή ε, του Προέδρου άρχισε η τρίτη φάση της κρίσης που είναι μια φάση αντίστασης, ένοπλης αντίστασης ε, η απόπειρα πραξικοπήματος τον Μάιο που απέτυχε βεβαίως ριζοστικοποίησε τις δύο πλευρές σκλήρινε την στάση της εξουσίας βεβαίως, αλλά σκλήρινε και τη στάση της αντιπολίτευσης και κυρίως ε, η επανεκλογή του Προέδρου Πουριπιζά το καλοκαίρι έδωσε την εντύπωση ε, και έθεσε τέλος στις απόπειρες μεσολάβησης της διεθνούς κοινότητας και έδωσε στην αντιπολίτευση την εντύπωση ότι υπήρχε μία μόνο επιλογή αλλαγής και ότι αυτή ήταν η ένοπλη αντίσταση. Βλέπουμε σε αυτή την τρίτη φάση της κρίσης στο Μπουρούντι ότι υπάρχει ε, μια διπλή κίνηση κλεισίματος ε, του καθεστώτος, ε, ένα κλείσιμο εσωτερικό αλλά και εξωτερικό που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Το κλείσιμο το εσωτερικό επισημάνθηκε με την εγκατάλειψη ορισμένων στελεχών της εξουσίας SM5-SNDD και η μετριοπαθής πτέρυγα έφυγε τώρα από το κόμμα και αυτό το κλείσιμο χαρακτηρίστηκε από την εγκατάλειψη πολλών μη κυβερνητικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που εξορίστηκαν όταν άρχισε η βία. Επίσης παρατηρούμε μια μεγάλη δυσπιστία της εξουσίας απέναντι στο στρατό και όπως είπε και η πρόεδρος στην εισαγωγή της έχουμε ένα τηλεσίγραφο από την εξουσία ε, στις συνοικίες ε, των ανταρτών με όρους που υπενθυμίζουν την ορολογία που χρησιμοποιείται το κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στο Μπουρούντι. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει σαφής απόσταση της εξουσίας ε, με την αρχή της ειρηνικής συνύπαρξης μεταξύ εθνοτήτων που καθιερώθηκε από τη Συμφωνία της Αρούσα το 2000 και που έθεσε τέρμα στον εμφύλιο πόλεμο. Βλέπουμε παράλληλα και με ένα κλείσιμο ε, εξωτερικό που χαρακτηρίζεται από ε, μία εναντίωση στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Πολλοί διεθνείς δημοσιογράφοι που πήγαν του τελευταίου μήνες ε, στο Μπουρούντι απειλήθηκαν, πολλοί ανταποκριτές τοπικοί ε, της, του διεθνούς τύπου δέχτηκαν επιθέσεις της αστυνομίας. Η κυβέρνηση ζήτησε την απομάκρυνση του πρέσβη του Βελγίου και επίσης κατηγόρησε το Βέλγιο και ότι βοηθάει την ε, αντιπολίτευση, την ένοπλη. Βλέπουμε ότι αναπτύσσεται ένας προφορικός πόλεμος ανάμεσα στη Μπουζουμπούρα και στο Κιγκάλι και μόνο ε, διάφορα μέτρα διακοσμητικά λήφθηκαν από την εξουσία ούτως ώστε να απαντήσει στα αιτήματα της διεθνούς κοινότητας όπως παραδείγματος χάρη η αναβολή για μερικές εβδομάδες των εκλογών. Αυτό που φοβίζει σήμερα τους πολίτες στο Μπουρούντι είναι ότι όλα τα γεγονότα που εξελίσσονται κυρίως από το μήνα Απρίλιο υπενθυμίζουν τα έτη που προηγήθηκαν του εμφυλίου πολέμου. Τα γεγονότα αυτά είναι παρόμοια, άρνηση του διαλόγου, κλείσιμο της πολιτικής σκηνής, καταπίεση, δολοφονίες στοχευμένες και όλα αυτά μας δείχνουν ότι επανέρχεται το παρελθόν και όλοι οι κάτοικοι του Μπουρούντι με τους οποίους συζητούμε το αναφέρουν αυτό, το επισημαίνουν αυτό, δηλαδή ότι αυτά που σημαίνουν εδώ και μερικούς, συμβαίνουν εδώ και μερικούς μήνες θυμίζουν τα όσα ε, συνέβησαν στην δεκαετία του 90 και οδήγησαν στον εμφύλιο πόλεμο. Υπάρχουν δύο ή τρία σενάρια επιτάπητος για τους επόμενους μήνες και που είναι ανησυχητικά. Το πρώτο σενάριο είναι βεβαίως αυτό μιας νέας απόπειρας πραξικοπήματος λόγω των εσωτερικών εντάσεων στις υπηρεσίες ασφαλείας. Το δεύτερο σενάριο είναι η ανάπτυξη μιας γκερίλας, ενός ανταρτοπόλεμου σε ορισμένες ζώνες της χώρας που θα τροφοδοτείται από την απομάκρυνση, από την εγκατάλειψη ορισμένων στρατιωτικών, από νέους, από την Μπουζουμπούρα και πρόσφυγες που τώρα ανέρχονται περίπου σε 207.000 πρόσφυγες σε 8 μήνες, δηλαδή μια ροή σημαντική ατόμων έφυγαν από το Μπουρούντι ε, και κατέφυγαν στην Τανζανία, στη Ρουάντα και στην Δημοκρατία του Κονγκό. Το άλλο σενάριο είναι μια καταπίεση βίαιη στις συνοικίες των ανταρτών ε, στην Μπουζουμπούρα με παράπλευρες ε, ε, ζημίες που θα έδιωχναν τους ε, αντιπολιτευόμενους από την πρωτεύουσα, αλλά δεν θα επέλυαν τίποτα, απλώς θα ενίσχυαν το σενάριο ενός ανταρτοπολέμου. Υπάρχει όμως και ένα στοιχείο θετικό. Δηλαδή έχουμε την εντύπωση ότι στο Μπουρούντι οι μάζες, ο λαός είναι πιο όριμος από την κυβέρνηση. Η εθνικιστική ρητορία της εξουσίας δεν πέτυχε, δεν είδαμε ε, διεθνωτικές διενέξεις και αντιπαραθέσεις. Δεν συμβαίνει αυτό. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν θα επισυμβούν, αλλά νομίζω ότι ο πληθυσμός είναι κάπως συγκρατημένος ε, και παίρνει τις αποστάσεις του σε σχέση με αυτήν την εθνοτικίστικη ε, ρητορία ορισμένων μελών της κυβερνήσεως που θέλουν να δώσουν την εντύπωση ότι αυτή η ανταρσία είναι μια εκδίκηση αυτών που έχασαν την εξουσία μετά τη συμφωνία της Αρούσα ε, και ότι ε, δεν αντιτίθενται στην τρίτη επανεκλογή του Προέδρου. Με τις περιστάσεις αυτές, η International Crisis Group ε, πιστεύει ότι υπάρχουν μέτρα που μπορούν να ληφθούν και διδάγματα να εξαχθούν. Οι στοχευμένες κυρώσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ενημερωθούν και ίσως να παραταθούν λόγω της εξέλιξης της κρατικής καταπίεσης. Εάν οι διαβουλεύσεις του άρθρου 96 δεν καταλήξουν, θα απαιτηθεί ε, να σκεφτούμε ε, μια διακοπή επιλεκτική της βοήθειας της Ευρωπαϊκής, εφόσον η βοήθεια ε, η ανθρωπιστική, η κοινωνική πρέπει να διαφυλαχθεί και να αυξηθεί, ενώ η θεσμική βοήθεια, η βοήθεια η δημοσιονομική θα πρέπει να ε, τερματιστεί, να ακυρωθεί. Θα πρέπει να περιλάβουμε τον Μπουρούντι στο διάλογο που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις γειτονικές χώρες, Τανζανία, Ρουάντα, Κένια, Ουγγάντα, και βεβαίως στην ε, δημοκρατία του Κονγκό. Μας φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ήδη επέδειξε ε, την υποστήριξη στις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον Μπουρούντι να εξακολουθήσει να τη στηρίζει σε ένα κλίμα όπου η ζωή τους κινδυνεύει πάρα πολύ συχνά και να υποστηρίξει μια εργασία ε, που θα καταπολεμήσει το κλείσιμο της χώρας στην πληροφόρηση. Θα πρέπει επίσης να, να διευκολυνθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτω ώστε να υπάρχουν συναντήσεις ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση με ένα πρόγραμμα που θα πρέπει και μια ατζέντα μια θεματολογία που θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή. Επίσης, η ανάπτυξη ε, των ε, παρατηρητών ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να υποστηριχθεί και να σκεφτεί κανείς τη συμμετοχή του στρατού του Μπουρούντι σε ειρηνευτικές διαδικασίες των οποίων ένα μέρος χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αμφισβητείται αυτή η συμμετοχή. Αυτή η κρίση δεν γεννήθηκε χτες, ορίμασε κατά τη δεύτερη θητεία του Προέδρου και αναδεικνύει ότι το θέμα της τρίτης θητείας που τίθεται στο Μπουρούντι και ε, στο Δημοκρατία του Κονγκό και στο Κονγκό Μπραζαβίλ και στην Κένια είναι ένα θέμα ε, το οποίο μπορεί ε, να επιφέρει νέες ταραχές σε όλη την περιοχή και θα πρέπει πολιτικά να αντιμετωπιστεί με πάρα πολύ σοφροσύνη και πάρα πολύ δεξιότητα και το Μπουρούντι είναι ένα προηγούμενο για όλες τις χώρες της περιοχής. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα δώσω πρώτα το λόγο σε δύο συναδέλφους που ζήτησαν το λόγο και μετά θα έχουμε και τον εκπρόσωπο της πρεσβείας του Μπουρούντι. Ο κύριος Μπένας Μέικερ πρώτα και μετά κύριε Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω Ολλανδικά. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την παρουσίαση που μας κάνατε. Οι εξελίξεις είναι πολύ ανησυχητικές. Πραγματικά μας αποτροπιάζουν και θεωρώ ότι αυτό μας φέρνει στο παρελθόν. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Οι διεθνείς παράγοντες θεωρούν ότι το Μπουρούντι είναι μια μικρή χώρα με μικρή επιρροή, με μικρή γεωπολιτική σημασία. Συνήθως λοιπόν τα τελευταία χρόνια στοχεύουμε περισσότερο και μας απασχολεί περισσότερο το Κονγκό, η Ρουάντα και κατά την άποψή μου αυτό είναι σφάλμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει σίγουρα να εξάγει κάποια διδάγματα. Έχουμε πάρει μέτρα, έχουμε επιβάλει περιορισμούς, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να κάνουμε και κάτι παραπάνω. Οι εξελίξεις στον Μπουρούντι είναι απειλή για την σταθερότητα της όλης περιοχής, για την ειρήνη στην περιοχή των μεγάλων λιμνών καθότι τα σύνορα δεν είναι καθόλου ασφαλή τα σύνορα του Μπουρούντι και υπάρχουν απειλές που μπορεί να μεταφερθούν σε υπόλοιπ, στις υπόλοιπες χώρες της περιοχής. Καταρχήν λοιπόν θα πρέπει να ξαναδούμε την αναπτυξιακή μας πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη χρηματοδοτούν ένα μεγάλο τμήμα του ετήσιου προπολογισμού του Μπουρούντι. Η χώρα μου, αλλά και η Γερμανία, και η Ολλανδία έχουν σταματήσει την αναπτυξιακή βοήθεια. Το ίδιο θα πρέπει να κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την άποψή μου, γιατί ένα πολύ μεγάλο τμήμα αυτής της αναπτυξιακής βοήθειας ουσιαστικά τροφοδοτεί την διαφθορά και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν στοχεύουμε κάποιους μηχανισμούς ανεξάρτητης προστασίας, τη διάκριση των εξουσιών, έτσι ώστε οι συμφωνίες αρούσαν να γίνουν σεβαστές. Όπως σας είπα, το Μπουρούντι βρίσκεται στην καρδιά της Αφρικής, στην περιοχή των μεγάλων λιμνών. Και η ερώτησή μου είναι αν δεν θεωρείται επικίνδυνο αυτές οι προσφυγικές ροές να κινητοποιήσουν και να τροφοδοτήσουν νέες εξεγέρσεις στη Ρουάντα και στις γύρω περιοχές. Τα γεγονότα στο Πουρούντι μήπως θα επηρεάσουν και τις εκλογές στη Ρουάντα του 2017. Η Ουγγάντα, εξ ονόματος των πέντε χωρών της Ανατολικής Αφρικής, προσπάθησε να παίξει ένα λόγο μεσολαβητή για να ξεπεραστεί η κρίση στον Μπουρούντι. Όμως διακόπηκαν ε, αυτές οι προσπάθειες και η ερώτησή μου είναι αν πιστεύετε ότι μπορεί η Ουγγάντα να συνεχίσει να παίζει ένα ρόλο εν μέσω αυτής της τρομοκρατίας και της βίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Εθνής Κοινότητα, αντιδρά σωστά κατά την άποψή σας. Και μία τελευταία ερώτηση, σύμφωνα με το άρθρο 96 της ε, Συμφωνίας Κοτονού, πρέπει να υπάρξει διαβούλευση 30 ημέρες μετά από μία πρόκληση. Έχει οριστεί κάποια ημερομηνία με τις αρχές του Μπουρούντι. Έχετε κάποιες πληροφορίες όσον αφορά αυτή τη διαβούλευση κυρία Κέγκε που είχε ζητήσει το λόγο, αλλά δεν την είχα δει. Ευχαριστώ. Ελένα. Θα ήθελα και εγώ να θέσω κάποιες ερωτήσεις, αλλά να κάνω και ένα σχόλιο. Γιατί η κρίση του Μπρούντι δεν είναι κάτι μεμονωμένο. Δυστυχώς είναι μια κρίση η οποία μπορεί να εμπλέξει όλη την περιοχή των Μεγαλυνών. Γι' αυτό σήμερα το να επιλύσουμε το ζήτημα του Μπουρούντι είναι ουσιαστική ε, σημασία για να μπορέσουμε να δώσουμε μία απάντηση σε όλες τις χώρες ε, που θα πάνε σε εκλογέ. εάν συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί ακριβώς αυτό είναι το ζήτημα. Αν ε, δεν αντιμετωπιστεί καλά το θέμα του Μπουρούντι, θα υπάρχουν συνέπειε σε όλες τις άλλες χώρε και νομίζω ότι θα δούμε το ίδιο σενάριο με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και εκτοπισμένους. Έτσι λοιπόν θα είναι καταστροφικές οι συνέπειες στον πληθυσμό. Και σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια εξουσία που μπορεί να ασκηθεί. Ε, πρέπει ουσιαστικά να δούμε και τις δηλώσεις που κάνει τις τελευταίες μέρες η κυβέρνηση του Μπουρούντι. Ουσιαστικά ορίζουν τις Βρυξέλλες ως ε, τους λομπίστες ε, του νέου απικισμού. Αυτές είναι δηλώσεις ε, που προέρχονται από την κυβέρνηση και εγώ τις καταδικάζω. Θα ήθελα να κάνω λοιπόν τώρα εδώ κάποιες σκέψεις. Θα πρέπει να ρωτήσουμε το εξής. Ε, πρέπει να ζητήσουμε να απελευθερωθούν αμέσως όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι, αλλά και οι δημοσιογράφοι και οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει να ζητήσουμε από το Μπουρούντι ε, το εξής. Αν δεν σεβαστεί τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης ΑΚΕ, ότι θα προβούμε σε διαβούλευση για το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και σε μια δημοκρατική λύση που θα πρέπει να γίνει αποδεκτή από όλους τους εμπλεκομένους. Δεν θα πρέπει να κάνουμε κάτι τέτοιο, ακόμη για να έχουμε την εξουσία, θα πρέπει να ζητήσουμε μία αποστολή παρατηρητών για το θέμα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εγώ θεωρώ ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο τον Μπουρούντι, αλλά την ευρύτερη περιοχή. Ευχαριστώ κυρία Μπέβερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι πιο επικριτική σήμερα, γιατί ε, η κριτική ε, δεν ε, κατευθύνεται μόνο στον Μπουρούντι, δεν μας εκπλήσει τόσο το γεγονός, αλλά είναι λυπηρό η κριτική μου είναι η εξή. Ε, Πόσε φορέ η Ευρωπαϊκή Ένωση πιάνεται ξαπίνη όταν συμβαίνει κάτι. Για μένα είναι δύσκολο να το κατανοήσω αυτό. Γιατί τα σημάδια, τουλάχιστον για το θέμα του Μπουρούντι, υπήρχαν εδώ και καιρό. Όχι μόνο από το 2014, αλλά από την αποστολή παρατήρηση των εκλογών το 2010. Θυμάμαι τότε όταν είχα θέσει μια ερώτηση σε σχέση με τους κινδύνους που υπάρχουν εκεί, μας είπαν «Ε, όχι, όχι, ο μόνος κίνδυνος είναι τα αυτοκινητιστικά δυστυχήματα. Και μεταξύ του πρώτου και δεύτερου γύρου των εκλογών είχαμε πάνω από 100 νεκρούς, είχαμε επιθέσεις με χειροβομβίδες συνέχεια και ούτε καν η αποστολή δεν μπόρεσε να εργαστεί και να συνεργαστεί με τους παρατηρητές που ήταν εκεί βραχυπρόθεσμα. Τώρα, κατόπιν όλων αυτών κάναμε μια αξιολόγηση για να δούμε τι έγινε εκεί. Και πιστεύω ότι η έλλειψη διαφάνειας σε ό,τι αφορά ορισμένα τμήματα της εκλογικής διαδικασίας ήταν ήδη κάτι εμφανές για μας και στο ότι θα έπρεπε να είμαστε ακόμη πιο προσεκτικοί για το θέμα του Μπουρούντι. Δυστυχώς τότε, κυρίως ο πρεσβευτής μας εκεί δεν ήθελε να δει την πραγματικότητα. Βέβαια άλλαξαν τα πράγματα, αλλά τότε υποστήριξη και από κάποιους πρέσβεις ήταν ε, δύσκολο να κατανοηθεί από δική μου πλευρά, κυρίω όταν βλέπαμε ότι πρόκειται για πολλά χρήματα, στέλνονταν πολλά χρήματα για να υποστηριχθεί μια χώρα η οποία είναι διαφθαρμένη ως το κόκαλο. Έτσι λοιπόν, εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί για το πώς κατανοούμε τη δική μας οικονομική βοήθεια δεν θέλουμε φυσικά να ενθαρρύνουμε και υποστηρίξουμε τη διαφθορά σε μια χώρα και δεν μιλώ μόνο για τον Μπουρούντι, αλλά για οποιαδήποτε χώρα. Εγώ συμφωνώ να υπάρχει άμεση στήριξη των ΜΚΟ ανθρώπων που πραγματικά χρειάζονται τη βοήθεια μας, αλλά όχι μέσω διεφθαρμένων κυβερνήσεων. Γιατί τα χρήματά μας πάνε στους δικούς τους λογαριασμούς ή στην τσέπη τους. Όμω, για τόσα συμβαίνουν τώρα στον Μπουρούντι, αναρωτιέμαι πράγματι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι η μόνη, δεν νομίζω ότι είναι η μόνη που πρέπει να κάνει κάτι. Θα πρέπει να συνεργαστεί και με την Αφρικανική Ένωση, γιατί θα πρέπει να εμπλακούμε ισχυρά στην ευρύτερη περιοχή. Και φυσικά και εγώ συμμερίζομαι τις ανησυχίες Κυρίω όταν μιλάμε για την ευρύτερη περιοχή των μεγάλων λιμνών. Ευχαριστώ κυρία Βέμπερ, η κυρία Γκόμε. Νομίζω ότι η δήλωση είναι πολύ σημαντική αυτή που μόλις ακούσαμε. Γιατί δυστυχώς η συμφωνία, αν θέλετε, της Κοτονού, η δική μας πολιτική, οι δηλώσεις μας και η πραγματικότητα, αν θέλετε, ο τρόπος που υλοποιούνται όλα αυτά, έχουν τεράστιες διαφορές. Και αυτό είναι ξεκάθαρο όταν κοιτάξει κανείς τι συμβαίνει στην Αφρική και στην περίπτωση του Πουρούντι. Αυτές οι αντιφάσεις και οι διαφορές είναι εμφανέστατες. Σήμερα δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αυτήν την κατάσταση. Σήμερα βλέπουμε ότι αυτή η αναπτυξιακή πολιτική ουσιαστικά καθοδηγείται από έναν τομέα ο οποίος δεν στηρίζει ούτε τον κόσμο, ούτε τα ανθρώπινα δικαιώματα, ούτε την ανάπτυξη τελικά. Βεβαίως πρέπει να έχουμε επαφή με τις αρχές των χωρών αυτών για να γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Πρέπει όμως να είμαστε και αποφασιστικοί όσον αφορά τον έλεγχο του πού πάει η βοήθεια αυτή, η χρηματοδότηση αυτή, αν πηγαίνει για τον εκδημοκρατισμό ή για την διαφθορά, για την ενίσχυση καθεστώτων που ενισχύουν αυτήν τη διαφθορά. Αυτό που είδατε εσείς στο Μπουρούντι το είδα εγώ το 2005 στην Αιθιοπία με παρόμοιες δυσκολίες και προκλήσεις. Η Σεσίλια μετά την Ιγυρία πήγε στο Μπουρούντι πολύ πρόσφατα και είναι τρομερή κατάσταση παρόλες τις απειλές της, βλέπουμε ότι οι χειρότερες ε, από τις σκέψεις μας, από τους φόβους μας, τελικά υλοποιήθηκαν, βγήκαν αληθινοί. Και βεβαίως υπάρχουν πολιτικοί κρατούμενοι, υπάρχουν θύματα, δολοφονίες. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, να αγνοούμε αυτά που συμβαίνουν και να μην επικρίνουμε τις αρχές μας γιατί ουσιαστικά στηρίζουν καθεστώτα τα οποία θέλουν απλώς να ενισχυθούν στην εξουσία και να παραμείνουν στην εξουσία. Δεν είναι δυνατόν, εγώ δεν στηρίζω αυτούς που λένε ότι πρέπει να συνεχίσουμε. Πρέπει να στείλουμε μια ξεκάθαρη, αν θέλετε, έκκληση, ένα σαφές μήνυμα προς αυτούς που μπορεί να δραστηριοποιηθούν στο Συμβουλίο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και σε κάθε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ δεν υποστηρίζω την διακοπή της βοήθειας. Πρέπει απλώς να την κατευθύνουμε σε αυτούς που την χρειάζονται, σε αυτούς που προσπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα θύματα. Ευχαριστώ. Λυπάμαι που δεν μπορέσα να ακούσω την παρέμβασή σας. Αλλά μπορώ να σας πω ότι παρακολουθώ εκ του σύνεγγυς όσα συμβαίνουν στον Μπουρούντι με αυτή την ανησυχία και την πικρία βλέπουμε ότι επαναλαμβάνεται η ιστορία. Σιγά σιγά βλέπουμε να γίνονται τέτοια πράγματα και πλέον ε, είναι πολύ δύσκολο να αντιδράσουμε για πρόληψη ούτε καν μιλάμε. Εγώ θα ήθελα να τονίσω το ψήφισμα των ΗΕ που θα ψηφιστεί το απόγευμα, υποθέτω ότι το αναφέρατε και είναι σημαντικό το Συμβούλιο Ασφαλείας να είναι αρκετά αποφασισμένο. Ξέρω ότι έχει τεθεί αυτό το θέμα και στην, ε, στις γαλλικές αρχές και από ό,τι φαίνεται έχει υπάρξει ε, μια αποδυνάμωση στις απαιτήσει. Όμως, ε, εγώ ελπίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να αντιδράσουμε και να οθήσουμε τα Ηνωμένα Έθνη να υιοθετήσουν αυτό το ψήφισμα. Και επίση, ε, για μια φορά να είμαστε και στη θέση να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μα για να επιβάλλουμε κυρώσει ή οι πόροι να φτάσουν στους δικαιούχους. Δεν θέλουμε οι πόροι να φτάνουν ε, στα χέρια ανθρώπων της κυβέρνησης που δολοφονούν ανθρώπους, ε, που μπλοκάρουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και που ασκούν ε, πολιτικές διώξεις εντελώς απαράδεκτες. Οι ουσιαστικά οδηγούν σε ένταση και ριζοσφαστικοποίηση της βίας. Άκουσα τι είπαν και οι συνάδελφοι. Εγώ πιστεύω ότι εδώ ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ενισχύσουμε αυτές τις δράσεις και πρέπει να συνεργαστούμε και με την Επιτροπή Ανάπτυξης και Ανθρωπιστικής Βοήθειας αλλά και με τα υπόλοιπα όργανα του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Μπεσέρα. Παρακαλώ αν θέλετε το λόγο τον έχετε πρόσωπο της Πρεσβείας του Μπουρούντι. Ευχαριστώ που μου ξαναδίνετε το λόγο κυρία Πρόεδρε. Άκουσα τις παρεμβάσεις ε, των διαφόρων ε, ομιλητών και μου φαίνεται ότι, ότι ε, μιλάτε για την κυβέρνηση του Μπουρούντι σαν να είναι ο μόνος υπέτειος για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όπως είπε ο πρώτος ομιλητής, είχαμε λοιπόν αυτήν την αντιπολίτευση από το 2015, την Αντερσία που αμφισβητεί την εκλογική διαδικασία και αυτή η κίνηση έγινε μια τρομοκρατική οργάνωση που έπειρε όμοιρους ορισμένους πολίτες ε, από την Μπουζουμπίρα, ε, κατέστρεψε ορισμένα κτίρια ακόμα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσης συνέλαβε άτομα απλώς ε, που τα γνώριζε ελάχιστα και στόχευσε πολιτικές και στρατιωτικές προσωπικότητες. Και όπως και άλλες χώρες, η κυβέρνηση ε, του Μπορούντι ε, προσπαθεί να αφοπλίσει αυτούς τους κακοποιούς και να εξασφαλίσει την ασφάλεια στο Μπορούντι, πράγμα που κάνει κάθε κυβέρνηση. Βέβαια, η κυβέρνηση ε, μετανοεί για τα σφάλματα και τις γκάφες που γίνονται, αλλά ο αφοπλισμός γίνεται με πολύ επαγγελματισμό και πολύ διαφάνεια. Και δράτω με τις ευκαιρίες αυτής για να ευχαριστήσω τις ευρωπαϊκές χώρες που ε, συνέβαλαν ε, στην εκπαίδευση των δυνάμεων ασφαλείας και της δημόσιας τάξης. Σχετικά με τις εθνοτικιστικές ομιλίες ορισμένων προσωπικότητων. Πρόσφατα ο αρχηγός του κράτους έκανε μια δήλωση για να διαβεβαιώσει τον πληθυσμό και την διεθνή κοινότητα ότι δεν θα υπάρξει ποτέ πόλεμος και γενοκτονία στο Μπουρούντι. Το μήνυμα της Δευτέρας ε, Νοεμβρίου επεξηγήθηκε από τις 8 Νοεμβρίου διότι υπήρξαν ερμηνείες εσφαλμένες διότι ένα μέρος ε, της ριζοσπαστικής ε, αντιπολίτευσης και κέντρα εξωτερικού παρερμήνευσαν τη δήλωση αυτή. Έχουμε ε, τα μέσα ε, ασφαλείας ε, τα οποία δίνουν λογαριασμό για την ασφάλεια της χώρας και τον αφοπλισμό αυτών που προσπαθούν να επιτεθούν σε θεσμούς που έχουν εκλεγεί δημοκρατικά. Τον Οκτώβριο του 2015 η έκθεση έλεγε ότι η κυβέρνηση είναι σίγουρη, εκτός, ε, έχει ασφάλεια εκτός από μια ε, συνοικία ε, στην Μπουζουμπούρα και είναι, παρέχει ασφάλεια στις 302 διαμερίσματα του Μπουρούντι. Γίνεται λόγος για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρξουν φυλακίσεις, υπάρχουν, αλλά οι φυλακίσεις γίνονται σύμφωνα με τον νόμο και δεν μπορούμε να απελευθερώσουμε έτσι φυλακισμένους, κρατούμενους χωρίς να έχουν δίκαστεί και αυτό πράττει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και υπάρχει μια Επιτροπή Δικαστικής Έρευνας που εξέφερε μια έκθεση σχετικά με τις, τη βία την προεκλογική και σε σχέση προσπαθήστε να κλείσετε, να τελειώσετε. Ναι, υπήρξε επίσης μια διαδικασία για το πραξικόπημα της 13ης Μαΐου και του υπέτειους και έχουμε μια Εθνική Επιτροπή Ανεξάρτητη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που ε, δημοσιεύει εκθέσεις τακτικά. Πρόσφατα το Μπουρούντι επελέγει ε, για να γίνει μέλος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Αυτά είναι καλά σημάδια το Μπουρούντι σέβεται τους, ε, τις διεθνείς συμφωνίες και τους νόμους όσον αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και νομίζω ότι στην περιοχή δεν είναι ο χειρότερος μαθητής. Και ε, οι παροτρύνσεις για κυρώσεις ε, και εναντίωση στην σημερινή εξουσία για να απομακρυνθεί δεν κάνει παρά να επιδεινώνει την κατάσταση. Κανείς δεν αναφέρθηκε στην ευθύνη των ανταρτών για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, δεν γίνεται λόγος για τις επιθέσεις κατά των αστυνομικών. Όλοι φωνάζουν για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά κανείς δεν μιλάει για το ότι πυροβολούνται οι αστυνομικοί. Θα πρέπει να είμαστε πιο επίοικείς και να ξέρουμε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη οι χώρες εταίροι του Μπορούντι θα πρέπει να εξακολουθήσουν να στηρίζουν τη χώρα ούτως ώστε η εσωτερικός διάλογος ή ο διάλογος με την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδώσει καρπούς, τους καρπούς που αναμένουμε όλοι. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Παντζέρη. είναι και απόσταση από τη χώρα που δεν μας βοηθά να εστιάσουμε στα προβλήματα. Όμως, ε, εμένα μου φαίνεται το πρόβλημα αρκετά απλό, παρόλη τη δραματική χρειά. Έχουμε παραβίαση των συμφωνιών της Αρούσα. Αυτό είναι το πρώτο δεδομένο. Κατά Κατόπιν έχουμε έναν ηγέτη, ο οποίος έχει γραπωθεί από την εξουσία και θέλει, παραβιάζοντας αυτές τις συμφωνίες, να εκτίσει και τρίτη αυτό είναι το κύριο πρόβλημα. Και η δική μου εντύπωση είναι ότι η σημερινή ε, πολιτική εξουσία στον Περούντι οδηγεί τη χώρα στην Άβυσσο. Έτσι λοιπόν θα ήθελα από τη μία πλευρά να υπάρξει μεγαλύτερη συνειδητοποίηση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της διεθνούς κοινότητας και ελπίζω το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών ε, να ε, προσεγγίσει απευθείας το πρόβλημα, ότι πρέπει δηλαδή να υπάρχει άμεση παρέμβαση, γιατί εγώ ανησυχώ ότι στον Περούντι μπορεί να επαναληφθούν τα όσα είδαμε στη Ρουάντα. Και το δεύτερο πολύ απλό στοιχείο, το είπαν και κάπω οι συνάδελφοι, εδώ, σε αυτή την επιτροπή, είναι εύκολα τα πράγματα. Όμως ε, σε ευρύτερη σύνθεση είναι πιο δυσκολία. Έχουμε τώρα την αναθεώρηση των συμφωνίων των κοντονιστών μέλλον και όταν μιλάμε για εμπορικές συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών θα ήθελα να υπάρχει μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ του σκέλους των ελεύθερων συναλλαγών και της αναπτυξιακής συνεργασίας. Ακόμη και αν ε, χρησιμοποιούμε στο δυνατόν καλύτερα τα όσα έχουμε ε, τώρα στη διάθεσή μας. Ε, πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή, όχι από την ουρά του ζητήματος και πρέπει να δούμε ακριβώς τις σχέσεις που έχουμε με όλες τις αφρικανικές χώρες και κυρίως αυτές που βρίσκονται σε κρίση. Ευχαριστώ. κύριε Βρυκούλο. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, το Μπουρούντι είναι ίσως περιφερειακό θέμα, το οποίο δεν μπορεί να λυθεί με περιφερειακά μέτρα. Η Νότια Αφρική από ό,τι φαίνεται δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το θέμα και δεν θέλει να συνεχίσει την προσπάθεια του Νέλσον Μαντέλα για την συνέχιση της συμφωνίας. Ξέρουμε ότι η όλη περιφερειακή προσπάθεια δεν ε, λειτουργεί με ενότητα. Υπάρχουν μέλη τα οποία έχουν πολύ συγκεκριμένες εκλογικές προκλήσεις, όπως ο πρόεδρος του Μπουρούντι και ο πρόεδρος της Ουγκάντα σαν μεσολαβητής σίγουρα δεν μπορεί να επιλύσει εκλογικά προβλήματα στον Μπουρούντι αφού ο ίδιος αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα στη χώρα του. Το άλλο θέμα που θίξατε, ότι δηλαδή υπήρχαν πολλές ενδείξεις ότι θα οδηγούμασταν σε αυτή την κρίση, ναι, υπήρξε μετά τις εκλογές του 2010 μια ολόκληρη καταστολή και περιορισμός ελευθερίας έκφρασης, η Συμφωνία Αρούσα με προβλήματα όπως παραδείγματος χάρη σε θέματα δικαιοσύνης, το θέμα του ποινικού δικαστηρίου, παραδείγματος χάρη που δεν θέλησε να υλοποιήσει η κυβέρνηση. Η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δράσει στο Μπουρούντι. Είναι ο πρώτος, αν θέλετε, χρηματοδότης. Ένα μεγάλο τμήμα του κρατικού προπολογισμού προέρχεται από εξωτερική χρηματοδότηση και αναπτυξιακή βοήθεια. Δεν πρέπει λοιπόν σε καμία περίπτωση να πολλαπλασιαστεί το ενδεικτικό εθνικό πρόγραμμα όπως έγινε το 2014, ενώ φαινόταν ότι θα υπέλθει εκλογική κρίση και βάσει του άρθρου 8 είδαμε ότι καμία συγκεκριμένη πρόοδος δεν μπορούσε να επιτευχθεί. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να εξισορροπηθεί η ευρωπαϊκή αναπτυξιακή βοήθεια με την έννοια ότι πρέπει να στηρίξουμε και την κοινωνία των πολιτών αλλά και τα θεσμικά όργανα. Στο εθνικό ενδεικτικό πρόγραμμα του 11ου ΦΕΔ διαπιστώνουμε ότι πρέπει να ξαναδεί κάποιο ε, τη στήριξη μια κυβέρνηση η οποία έχει αρχίσει να σκληραίνει σημαντικά τη στάση της. Οι αρχές του Μπουρούντι έκαναν ακριβώς το αντίθετο από αυτό που ζητούσαν οι διεθνείς εταίροι για την ε, μεταρρύθμιση παραδείγματο χάρη ε, των δυνάμεων ασφαλεία, της αστυνομίας, παραδείγματο χάρη έκανε ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή σκλήρινε τη στάση της και στρατικοποίησε την αστυνομία αντί να κάνει το αντίθετο. Τώρα, τι διεθνή μέσα διαθέτουμε, διαθέτει η Διεθνής Κοινότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο Ασφαλείας, το οποίο αναφέραμε για ένα ψήφισμα, το οποίο προετοιμάζεται, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο είναι έτοιμο να ξεκινήσει έρευνες για εγκλήματα τα οποία εμπίπτουν τη αρμοδιότητά της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σαφώς και θα πρέπει να στηρίξει όλες αυτές τις προσεγγίσεις που έχει ξεκινήσει και τις προσπάθειες που έχει ξεκινήσει ο Γενικός Αγγελέας του Ποινικού Δικαστηρίου. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε τη συζήτησή μας για τον Μπουρούντι. Και βεβαίως υπενθυμίζω ότι για το άρθρο 96 της Συμφωνίας Κοτονού έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις, τουλάχιστον ζητήσαμε από τον Μπουρούντι να το κάνει στις 26 Οκτωβρίου. Στις 26 Νοεμβρίου ελπίζω 30 μέρες μετά να υπάρξει ανταπόκριση σε αυτό το αίτημα. Λοιπόν, τώρα συνεχίζουμε με τα όσα έχουν απομείνει στην μισή διάταξη. Ευχαριστούμε τον κύριο Βερκούλο να δούμε τώρα τι θα κάνουμε γιατί δεν έχουμε χρόνο και έχουμε τρία ζητήματα να συζητήσουμε. Και καθώς έχουμε καθυστερήσει, ο κύριος ε, Μάουρα και ο έχουν έρθει για να κάνουν ε, την ενημέρωση για τη Βενεζουέλα. Επομένω, ας ξεκινήσουμε από τη Βενεζουέλα, γιατί έχουμε εδώ τους συναδέλφους ε, που έχουν έρθει. Δυστυχώς δεν τα πήγαμε καθόλου καλά με το χρόνο σήμερα το πρωί. Όταν θέλετε παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόκειται για μια συζήτηση και κλεισμένων των θυρών. Δηλαδή, όσοι δεν είναι μέλη του Κοινοβουλίου ή εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων, θα πρέπει να εγκαταλείψουν την αίθουσα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Αλλά από ό,τι φαίνεται αυτοί είναι οι κανόνες και πρέπει να τους σεβαστούμε. Παρακαλώ όμως, επειδή δεν έχουμε χρόνο, όσοι πρέπει να αποχωρήσετε, να το κάνετε γρήγορα και με ησυχία. Por favor, please.